Παρακαλώ συνάδελφοι. Παρακαλώ, θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε την κοινή ακρόαση των τριών επιτροπών της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Επιτροπής Βιομηχανίας και Επιτροπής Γεωργίας. Εκ μέρους και των τριών επιτροπών, Έμβια, Άγκρη και Ήτρε, θα ήθελα να καλωσορίσω τους ε, εκπροσώπους καταρχήν των δύο άλλων επιτροπών, την κυρία Μια Πέτρα Κούπουλα Νάτρη από την Επιτροπή Ήτρε που θα προεδρεύσει στο δεύτερο τμήμα της ακρόασης και να καλωσορίσω και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, τον κύριο Πάβελ Πότς, αντιπρόεδρο της Ανλόγου Επιτροπής, που δεν ήρθε όμως μάλλον ακόμη. Όπως ξέρετε, η στρατηγική για τα δάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνει ένα πλαίσιο για τα θέματα των δασών και προτείνει ένας, μια συνεκτική και σφαιρική αντίληψη της διαχείρισης των δασών που καλύπτει τα πολλαπλά ωφέλη ε, των δασών και καλύπτει όλη την αλυσίδα αξία του δάσους. Και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2015 έκρινε ψήφισμα για τη στρατηγική των δασών με έμφαση στην ιδιαίτερη σημασία, την κρίσιμη σημασία που έχει μια αηφόρος διαχείριση των δασών και την τον πολυσχεδί οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό ρόλο των δασών και ε, ζητήσαμε την εξασφάλιση καλύτερου συντονισμού των τομεακών πολιτικών που άμεσα ή έμεσα συνδέονται με τη δασοκομεία. Το Σεπτέμβριο μάλιστα το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το πολιετές εφαρμοστικό της σχέδιο ως μέσο για την εφαρμογή της στρατηγικής για τα δάση με ε, συγκεκριμένο κατάλογο δράσεων για την περίοδο 2015-2020 με πρόβλεψη για μια αξιολόγηση που θα γίνει της στρατηγικής αυτής κατά το 2018. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να να εκτιμήσουμε την πρόοδο κατά την εφαρμογή αυτής της δασικής στρατηγική, υπό το φω και των νέων ε, ε, προκλήσεων στα πλαίσια και του πλαισίου κλίματος και ενέργειας του 2030, στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, της βιοοικονομίας, της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και του προβληματισμού μας για το μέλλον της κοινή γεωρικής πολιτικής και τις ανάγκες να ενισχύσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές. Γιατί είναι ένα θέμα οριζόντιο και ξέρουμε ότι τα δάση δεν είναι μόνο πολύ σημαντική πρώτη ύλη, αλλά διαδραματίζουν κέριο ρόλο στη βιοπικιλότητα και προσφέρουν και πολλές άλλες υπηρεσίες. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι πολυσχηδής και πολυεπίπεδος ο ρόλος ε, των δασών και της δασοπονίας. Σήμερα θα κάνω μια ανάλυση αυτής της ε, κατάστασης και γι' αυτό θα χωρίσουμε τη δημόσια μας ακρόαση σε τρία τμήματα. Αυτό έγινε με τη βοήθεια το, των γραμματιών των τριών επιτροπών. Το πρώτο τμήμα της ε, δημόσιας ακρόασης θα, το προεδρεύσει υποφαινόμενος, το δεύτερο εκπρόσωπο της Επιτροπής Ήτρια και το τρίτο εκπρόσωπο της Επιτροπής ΕΜΒΗ. Σε κάθε τμήμα θα έχουμε δύο σύντομες παρουσιάσεις. Γι' αυτό θέρμο παρακαλώ και απευθύνω έκκληση και στους καλεσμένους μας ε, να μην ξεπεράσουν το οκτάλεπτο που δικαιούνται για τις παρουσιάσεις τους. Επίσης, έκκληση προς τα μέλη των τριών επιτροπών ε, να τηρήσουν το ένα λεπτό που θα έχουν στη διάθεσή τους για την υποβολή των ερωτήσεων στους καλεσμένους εμπειρογνώμονές μας. Έχουμε περιορισμένο χρόνο για τη διεξαγωγή αυτή τη ακρόαση, γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί στην τήρησή του. Θα δώσω όμω πρώτο το λόγο στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην εκπρόσωπο συγκεκριμένα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Γιωζεφίν Λορίτ Χόφμαν, που είναι διευθυντή Αγροτικής Ανάπτυξης στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, που θα μας παρουσιάσει συντομία ε, την κατάσταση της σημερινής Ευρωπαϊκής Δασικής ε, Στρατηγικής και τις τελευταίες εξελίξεις ε, και τις προοπτικές. Κατόπιν θα περάσουμε στο πρώτο θεματικό τμήμα της ε, δημόσιας ακρόασης. Δεν θα κάνω λεπτομεριακέ παρουσιάσει για να μην χάνουμε χρόνο. Ευχαριστώ και πάλι και καλωσορίζω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ε, καλεσμένους μας εμπειρογνώμονες. Ε, και παρακαλώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι και αυτή αυστηρή στην τήρηση του χρόνου. Ένα δεκάλεπτο το πολύ. Έτσι έχουμε κρίνει με σκόπιμο τον επιμερισμό του χρόνου. Παρακαλώ δέκα λεπτά και όχι παραπάνω, αν γίνεται, κυρία Χόφμαν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα Καλησπέρα σε όλους κυρίες και κύριοι. Πρώτα θα ήθελα να εκφράσω, να σας μεταφέρω τα χαιρετήματα από τον Επιτροπό μου, ο δυστυχώς δεν μπορεί να παρευρεθεί στη σημαντική σημερινή συνεδρίαση. Αλλά εκ μέρους του θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τα μέλη του Κοινοβουλίου για το συνεχόμενο ενδιαφέρον που δείχνουν για την ε, στρατηγική. καθώς έχουμε τρεις σημαντικές επιτροπές που συζητούν το ζήτημα σήμερα. Πριν από ένα χρόνο, ο Επίτροπος Χόγκαν ήρθε στην κοινή συνεδρία των τριών επιτροπών για να έχει την πρώτη ανταλλαγή απόψεων με εσά και θα εστιάσω στο τι έχει συμβεί από τότε μέχρι τώρα και ποιε είναι οι ερχόμενες δράσει σε αυτό το τομέα. Τον τελευταίο χρόνο οι πολιτικέ σε σχέση με τη νοσοκομεία αποτελούν ένα κομμάτι Τη ευρωπαϊκή πολιτική γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση στα προϊόντα ε, τη νοσοκομεία και ξυλία. Και υπάρχουν πρωτοβουλίε σχετικέ με τη δασοκομεία, ειδικά αυτέ που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, το κλίμα, το περιβάλλον και την καινοτομία. Θα ξεκινήσω ωστόσο από το πιο δυσάρεστο γεγονό αυτό το χρόνο και είναι οι πυρκαγιέ που ήταν ιδιαίτερα σοβαρές, χωρίς προηγούμενο και που έθεσαν στο πρωτοσέλιδα, έφεραν στο πρωτοσέλιδα την, τα δάση μας. Είχαμε πολύ σοβαρές ζημιές στα δάση, αλλά αυτό που είναι ακόμα πιο σημαντικό και πιο θλιβερό είναι το γεγονός ότι είχαμε και θύματα ανθρωπινά θύματα στις ε, πυρκαγιές αυτές. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω τα συλληπιτήρια από τις οικογένειες των θυμάτων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει τα κρατη να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προκαλούνται από τον κίνδυνο πυρκαγιών και άλλων ακραίων φαινομένων, παρέχοντας ε, βοήθεια στην πυροσβεστική, σε πολιτικές αποκατάστασης και σε προγράμματα πρόληψης στο πλαίσιο της κοινή γεωργικής πολιτικής, αλλά και μέσω του ε, Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, της Περιφερειακής Πολιτικής των Πληροφορικών ε, Συστημάτων για τα περιβαλλοντικά προγράμματα. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική ως κομμάτι της ε, ε, γεωργικής προ... πολιτικής, το διάστημα αυτό το 2014 2020 το ποσό ανέρχεται στα 2,4 δισεκατομμύριο και το 70% αυτού του ποσού ε, κατανέμεται σε προμηθευτικά μέτρα μέτρα και στην αποκατάσταση. Αυτά αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι της ε, ε, αντιμετώπισης ε, ακραίων φαινομένων. Μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του έτους αυτού, η Επιτροπή ξεκίνησε διάλογο για το αν χρειάζεται περαιτέρω δράση από την πλευρά της συγκεκριμένα στην ενίσχυση της πρόληψης εν ώψη της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της οι δράσεις συμπεριλαμβάνουν μία ε, σύνοδο στην ε, Πορτογαλία το Φεβρουάριο και μία πρόταση από την Επιτροπή για τη δημιουργία ε, ένα εφεδρικό σώμα. Το 2003 η νομοθεσία που εγκρίθηκε σχετικά με την ε, βιωσιμότητα βασίζεται και στην ε, αρχή της ε, επικουρικότητας. Έχουμε ένα νέο σχέδιο δράσης στη στρατηγική αυτή και θα ήθελα στο μία να αναφερθώ στις 7, στους 7 τομείς να σας πω ποια είναι η κατάσταση. Πρώτα θα αναφερθώ στην ε, βιώσιμη διαχείριση υπό την ε, κοινωνική πολιτική. Υποστηρίζουμε τις κοινότητες της υπαίθρου στην προσπάθειά τους να ε, φέρουν τις τομικές αλλαγές που χρειάζονται στα μέτρα σε σχέση με τα δάση. Αυτό που προβλέπονται για τα κράτη-μέλη ανέρχονται σε πάνω από 7 ε, εκατομμύρια ευρώ δημόσιων δεπανών στην περίοδο 2014-2020. Η εφαρμογή θα προσφέρει 500.000 εκτάρια δάσους, 70.000 εκτάρια ε, δασοκομείας και 4.000 ε, σε σχέση με το Natura και άλλο ένα και άλλα χιλιά 1,4 εκατομμύρια. Έχουμε επανέλθει στα επίπεδα προκρίσης και αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για τον τομέα. Η συνεκτική ε, δημιουργία κριτηρίων για την ε, βιοενέργεια θα συμβάλλει στην βελτίωση των επενδύσεων στον τομέα, παρέχοντας επαρκή ασφάλεια για τον τρόπο που ε, θα παράγεται η βιομάζα και πώς θα φτάνει στους καταναλωτές. όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και την πρόληψη των ε, πυρκαγιών. Η καλή διαχείριση συμβάλλει στην ευρωπαϊκή πολιτική ε, προσεγγίζοντας τους ε, στόχους για την παραγωγή καινοτόμων και βιώσιμων προϊόντων. Στην τελευταία συμφωνία του Παρισίου η Συμφωνία για την Αλλαγή Χρήσης Γης κάνει αναφορά για πρώτη φορά στα δάση και ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την, ε, στην κλιματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη πλευρά, τα δάση είναι πολύ ευάλωτα στις αλλαγές αυτές και η ευρωπαϊκή πολιτική για τα δάση ενθαρρύνει τις ε, επενδύσεις για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Η προστασία των δασών και του οικοσυστήματος και οι υπηρεσίες ειδικέ απαιτούν ως προτεραιότητα την ε, βελτίωση της εφαρμογής ε, της ε, οδηγίας Nature το τρέχον σχέδιο δράσης είναι η απάντηση της Επιτροπής σε αυτή την πρόκληση. Θα ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ φύσης, οικονομίας και κοινωνίας και είναι σχετικές με οι δράσεις με τα δάση. Οι καινοτόμε δράσεις και τα προϊόντα προωθούνται μέσω προγραμμάτων εντός ε, του σχεδίου ε, δράσης ε, καινοτομίας και στις ε, νέες επιχειρήσεις ε, για την βιοενέργεια συμπεριλαμβάνει και καταλήγουμε ότι η στρατηγική έχει κινητοποιήσει ιδιωτικές και δημόσιες ε, επενδύσεις, αλλά μπορεί να γίνουν περισσότερα στη διεύρυνση της αγοράς ε, για σχετικά προϊόντα. Έγινε μια αναθεώρηση της στρατηγικής και αυτό βοήθησε στο να γεφυρώσουμε τα χάσματα όσον αφορά τη συζήτηση και την εξέλιξη της ε, πολιτικής για τα δάση και την χρήση τους από τους εμπειρογνώμονες και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή είναι ένα πολύ σημαντικό φόρουμ για τη συντονισμό των ε, διαλόγων μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών σε όλα τα σχετικά με τα δάση θέματα. Όπως γνωρίζετε, αυτή η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τι εξελίξεις στην ε, βιοοικονομία, βιοποικιλότητα και τις σχετικέ πολιτικές και συνεργάζεται με άλλα τομεακά φόρουμ. Αυτή η Επιτροπή Σε αυτήν συμμετέχουν ε, και ενδιαφέροντα μέρη στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου και από την ε, δοσκομική μηχανία. Χθε είχαμε συνεδρίσει των δύο ομάδων της ε, ε, Μόνιμης Δασικής Επιτροπής, όπου συζητήθηκε η στρατηγική. Τελευταίο σημείο είναι να δούμε το, τα δάση από μια παγκόσμια προπτική, να δούμε τα διεθνή, τις πρωτοβουλίες, καθώς και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Νόμου από τις κυβερνήσεις που πετυχαίνει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Επιπλέον, ασχολούμαστε με την πρόθεση της ε, διαχείρισης, εφόρου διαχείρισης των δασών μέσω του Forest Europe και σε άλλα φόρουμ. Με άλλα λόγια, η Επιτροπή συνεργάζεται συχνά για να φέρει αποτελέσματα και είναι δεσμευμένη σε αυτές τις αρχές και ε, τους στόχους της στρατηγικής που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόλις τώρα ξεκινάμε την αξιολόγηση της εφαρμογής της στρατηγικής και σχεδιάζουμε να έχουμε τα αποτελέσματα διαθέσιμα τον επόμενο χρόνο, δηλαδή το 2018 θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε δράσεις και προτεραιότητες στη δεύτερη φάση του πολιτού ε, σχεδίου εφαρμογή να εντοπίσουμε κενά και ανάγκες ε, υπό το φως των νέων αναγκών ε, σε σχέση με τα δράση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Χόφμαν. Περνάμε στην πρώτη θεματική ενότητα της ε, δημόσιας ακρόασής μας που θα ασχοληθεί με την Ευρωπαϊκή Δασική Διακυβέρνηση, τη δασοπονία και τον ε, τομέα της ε, αγροτικής ανάπτυξης που στηρίζεται στο δάσος. Έχουμε ως πρώτο εμπειρογνώμονα τον κύριο Μάρκ Παλαχή, που είναι διευθυντής του Ευρωπαϊκού Δασικού Ινστιτούτου και εμπειρογνώμων στα θέματα του δάσους. Πρόκειται για μια διεθνή οργάνωση που δραστηριοποιείται έντονα σε αυτά τα θέματα τα δασικά και ο δεύτερος καλεσμένος μας στο, στην πρώτη ενότητα της ακρόασης είναι ο κύριος Χέικι Γκρανχόλμ από το Φιλανδικό Υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομεία με πολύχρονη πείρα στα θέματα της δασοκονίας και, ε, και μάλιστα μεταξύ άλλων είναι και συμπρόεδρος τη Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασία για την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Δασική Στρατηγική και συμπρόεδρος του Συμβουλίου ε, και Μέλλον ε, του Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα, για τα δάση. Από 8 λεπτά λοιπόν θα έχει ο κάθε καλεσμένος μας. Πρώτα το λόγο, το λόγο έχει ο κύριος Μάρκ Παλαχή. Ευχαριστώ πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Στη σύντομη εισήγησή μου θα ήθελα να μεταφέρω κάποιες σκέψεις και κάποια δεδομένα για τη σημασία των ευρωπαϊκών δασών ως χώρο για την βιώσιμη ανάπτυξη και θα ξεκινήσω με τον κύριο ρόλο μετασχηματισμού των δασό μα για την αλλαγή ενό ε, για την λογική δημιουργία ενό νέου οικονομικού μοντέλου το οποίο χρειαζόμαστε επιγόντω στα πλαίσια του, της βιωσιμότητας του πλανήτη. Κάτι το οποίο ως παράδειγμα, ως υπόδειγμα θα βασίζεται στην ανανεώσιμη ενέργεια ε, ως βάση της βιώσιμης οικονομίας και όπου η βιοοικονομία θα αποτελέσει την γεννητήρια δύναμη για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Οι βιολογικοί λοιπόν πόροι όπως ε, τα δάση και η βιοοικονομία είναι λοιπόν η βάση μιας βιώσιμης οικονομίας. Ε, εν τω μεταξύ όμως χρειαζόμαστε στο τομέα της ενέργειας μέχρι την αποανθρακοποίηση να δημιουργήσουμε διάφορα υλικά που θα αφορούν τι ε, συσκευασίε, μεταφορέ κτλ. Και αυτά τα υλικά θα πρέπει ακόμα να βασίζονται, να στηρίζονται στον άνθρακα. Θα πρέπει λοιπόν εντωμεταξύ να αντιμετωπίσουμε για το θέμα τη κλιματική αλλαγή. Οπότε αυτά τα υλικά που βασίζονται στον άνθρακα θα πρέπει να προέρχονται από κυρίω βιολογικέ πηγέ, πηγέ ανανεώσιμε, οι οποίε δεν περιέχουν καταρχά άνθρακα. Για να πετύχουμε όμω στην βιοοικονομία, θα πρέπει όχι μόνο να επικεντρωθούμε στην αντικατάσταση των ορυκτών πηγών μέσω ανανεώσιμων πηγών, αλλά θα πρέπει να δώσουμε στην οικονομία αυτή την ευκαιρία να αντιμετωπίσει τη δικασία αυτή ως μια αξιοποίηση της φύσης. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι η οικονομία μας επιτρέπει να οικοδομήσουμε μια, ε, μια σχέση συνεργασίας μεταξύ οικονομίας και οικολογίας. Και σε αυτό το πλαίσιο τα δάση έχουν ένα τεράστιο δυναμικό και θα πρέπει να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο όσον αφορά την δημιουργία μια βιώσιμη οικονομία, μια βιοοικονομία. Να σα εξηγήσω γιατί καταρχά τα ευρωπαϊκά δάση αποτελούν την κυριότερη υποδομή, τη βιολογική υποδομή του πλανήτη μα. Όχι μόνο επειδή καλύπτουν γύρω στο 40% τη επικράτεια Ένωση, αλλά επειδή αποτελούν το, τη μεγαλύτερη λεκάνη καταβόθρα διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή στην ουσία τα δάση μας είναι απαραίτητα για την ανθεκτικότητα των υπαίθριων και των αστικών κοινοτήτων, επειδή ακριβώς ε, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη δημιουργία πόρων, τα οποία, ε, πόρων οι οποίοι υποστηρίζουν την ε, βιωσιμότητα. Τα δάση μας όμως διαδραματίζουν και άλλο ένα σημαντικό ρόλο. Δηλαδή τα δάση μας τα οποία διαχειρίζονται αποτελούν την κύρια πηγή πόρων ανανεώσιμων που συνδέονται με τις ε, κατάλληλες ε, τεχνολογίες και μπορούν να μετα, μετατραπούν σε υλικά όπως το βαμβάκι και άλλα, τα οποία θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τα ορυκτά προϊόντα και να τα ξεπεράσουν ε, περιβαλλοντικά στους, ε, στους βιομηχανικούς τομείς, όπως τα πλαστικά, η οικοδομή κτλ. Οπότε αυτός ο τομέας λοιπόν βασίζεται στα δάση, παρουσιάζει ένα τεράστιο δυναμικό όσον αφορά την, με, τον μετασχηματισμό όλου αυτού του κλάδου σε σχέση με την κακή οικονομία. Τα δάση όμω και ο κλάδο των δασών δεν αποτελεί μόνο μια μελλοντική υπόσχεση, αποτελεί ήδη μια σημαντική οικονομική πραγματικότητα. Καμιά φορά υποτιμάται, αλλά θα δείτε εδώ στον πίνακα ότι οι βιομηχανίες που βασίζονται στα δάση έχουν μεγαλύτερη οικονομική κλίμακα από οποιοδήποτε άλλο βιομηχανικό κλάδο στους ε, τομείς του χάλιβα, των πλαστικών κτλ. Επιπλέον, τα δάση προσφέρουν πάνω από 3 εκατομμύρια θέσεις εργασία σε πάνω από 300.000 επιχειρήσεις, το οποίο είναι απαραίτητο για να έχουμε περιεκτική ανάπτυξη. Στην ουσία, λοιπόν, η, τα δάση παρέχουν τεράστιες ευκαιρίες για την κατανομή του πλούτου, των θέσεων εργασία, των υποδομών και των επενδύσεων σε όλες τις περιοχές της υπεθρία μας. Θα ήθελα όμως επίσης να τονίσω ότι θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι μιλητής, ότι τα δάση δεν είναι μόνο σημαντικά για να στηρίξουμε τις υπαίθριες περιοχές, είναι και κρίσιμα για την ανάπτυξη βιώσιμων πόλεων. Για ποιο λόγο. Διότι το ξύλο είναι το μόνο υλικό κατασκευή το οποίο είναι βιώσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με, τον κατάλληλο και, με κατάλληλους και αποτελεσματικούς τρόπους να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Στην ουσία δηλαδή αντικαθιστώντας ε, το τσιμέντο και το σίδηρο και το χάλιβα μειώνουμε κατά 50% το αποτύπωμά μας. Αυτό έχει τεράστια σημασία αν λάβετε υπόψη σας ότι ο τομέας της οικοδομής στην Ευρώπη και η οικοδομή αντιπροσωπεύει το 35% των ρήπων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο μείνουμε και τις ανάγκες θέρμασης και ψήξης. Για αυτούς, λοιπόν, για αυτούς τους λόγους τα δάση θα αποτελέσουν την ραχοκο... ραχοκοκαλιά των μελλοντικών αποτελεσματικών περιβαλλοντικά πόλεων. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν τονίζουμε τη σημασία των δασών μας και το δυναμικό τους ω πηγή, μελλοντική πηγή βιώσιμη ανάπτυξη. Όμως, για να διασφαλιστεί αυτό και να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή με την ανθεκτικότητα, θα πρέπει επιγόντως να αναπτύξουμε μια ολιστική και μακρόπνοη πολιτική και το αντίστοιχο πλαίσιο, ώστε να δώσουμε τα κατάλληλα κίνητρα και να προσελκύσουμε τις σωστές επενδύσεις για την διαχείριση ακριβώς, τη σωστή διαχείριση των δασών και δημιουργία ενός ενάρετου κύκλου, ο οποίος θα βασίζεται ακριβώς στην βιωσιμότητα, στην ανθεκτικότητα και στην ε, ε, βιοοικονομία. Αυτό αποτελεί μια προϋπόθεση για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Οπότε, στα πλαίσια ήδη αυτού που ανέφερα, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάση αποτελεί ένα πολύ συνεκτικό και αποδοσματικό εργαλείο το οποίο συνδυάζει προοπτικές και στόχους. Όμως αυτό δεν είναι το κύριο ζήτημα. Το κύριο ζήτημα, κατά την άποψή μου, είναι ότι αν η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωση για τα δάση αποτελεί μια, ένα στρατηγικό σημείο αναφοράς για την χάραξη άλλων παράλληλων πολιτικών. Ισχύει αυτό, συμβαίνει αυτό και αν όχι, για ποιο λόγο και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ώστε ακριβώς να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτή την σωστή στρατηγική. Θα ήθελα να καταλήξω τονίζοντας την ανάγκη για μια αποτελεσματική επιστημονική πολιτική. Μαζί με τη χάραξη της πολιτικής και την εφαρμογή της ε, στατικής της Ένωσης για τα δάση. Αυτή η διάδραση λοιπόν αυτών των στοιχείων θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην στρατηγική της Ένωσης για τα δάση και στην ισχύουσα δομή διαχείρισή του. Χωρί μια ισχυρή επιστημονική πολιτική και διάδραση δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά την ευρωπαϊκή πολιτική για τα δάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Παλαχή, ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σα, και επίση και τηρήσατε το χρόνο σα. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Χέικη Γκράνχολμ Παρακαλώ. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα τις τρεις επιτροπές σας για τη διοργάνωση αυτής της δημόσιας ακρόασης. Είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα ε, και περίτρανη απόδειξη του ζωηρού ενδιαφέροντος που έδειξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα θέματα της πολιτικής για τα δάση. Και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω την εμπειρία που έχουμε από πρώτο χέρι κατά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Δασικής Στρατηγικής μετά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής της. Ποια είναι τα βασικά μου μηνύματα. Πρώτον, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δάση είναι ένα πολύ καλό έγγραφο. Βέβαια, οι ζωτικές προτεραιότητες και προκλήσεις παραμένουν. Πώς θα ενισχύσουμε τη συνοχή και το συντονισμό κατά την προετοιμασία και την εφαρμογή της πολιτικής. Όπω επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή Δασική Στρατηγική, θα ήθελα και εγώ να τονίσω ότι τα δάση και η βιώσιμη δασική στρατηγική είναι συνδετικά στοιχεία και γέφυρε μεταξύ των αγροτικών, αστικών, βιομηχανικών και άλλων ε, οικοσυστημάτων και θα πρέπει να δούμε και τη, την κλίμακα, θα είναι περιφερειακή, τοπική, εθνική ή παγκόσμια. Πάντως υπάρχει δυνατότητα και ταυτόχρονα επιτακτική ανάγκη της βελτίωσης της εφαρμογής της ε, δασικής στρατηγικής. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην προετοιμασία της πολιτικής, στην εφαρμογή, καθώς και στην αξιολόγηση και την αναθεώρηση αν χρειάζεται. Ε, σε ποιον απευθύνεται η, στρατηγική των δασών, στη γενική, ε, στις Γενικές Διευθύνσεις Επιτροπής, στα κράτη-μέλη, στο Κοινοβούλιο, στη μόνιμη Επιτροπή για τα Δάση και άλλες ομάδες και ε, παράγοντες που συμμετέχουν στην εφαρμογή αυτής της δασικής πολιτικής. Και ποιος είναι ο μελλοντικός δρόμος, είναι, περνάει από την αντίληψη ότι τα δάση είναι τμήμα της λύσης και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική των Δασών να συνεχίζει να αποδίδει έργο και να αποφέρει καρπούς. Θα πρέπει τα θέματα των δασών να παραμείνουν υψηλή προτεραιότητα του προγράμματός μας και μετά το 2019-2020 και θα θέλαμε τα δασικά ζητήματα να συμπεριλαμβάνονται και στο νέο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και στο μελλοντικό νομοθετικό έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι έχουμε πολλά θετικά παραδείγματα και επιτεύγματα. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομεριακή αναφορά τους. θα σας μοιράσω και τις διαφάνειές μου. Ε, η εκπρόσωπος της Επιτροπής για την εφαρμογή αυτής της δεσικής στρατηγικής μας τόνισε μερικά από τα επιτεύγματα. Εδώ θα ήθελα να ε, τονίσω την συνοχή άλλων πολιτικών και μέσων, όπως είναι της αγροτικής ανάπτυξης, βιοποικιλότητας, βιοοικονομίας, τη επιβολή δασική νομοθεσία για κυβέρνηση και εμπορίου, φλεκτ και ούτω, ούτω καθεξής. Επίσης, ε, είχαμε ε, πολλές ε, χρήσιμες μελέτες που έγιναν στα πλαίσια της εφαρμογής, αλλά σε μερικέ περιπτώσεις ανακύπτει το ερώτημα ποια ήταν η αποτελεσματικότητα αυτών των μελετών για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Δάση. Οι εμπειρίες μας από την ε, εφαρμογή Κατά τη γνώμη μας, τα πιο θετικά παραδείγματα είναι αυτά στα οποία, για τα οποία συνεργαστήκαμε και η όλη προετοιμασία της στρατηγικής έγινε από κοινού ε, με τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για παράδειγμα, η ομάδα εργασίας ε, που ε, αξιολόγησε τα κριτήρια της βιώσιμης δεσικής στρατηγικής και το πώς εφαρμόζεται στα διάφορα, στις διάφορες πολιτικές, άσχετα από την τελική χρήση της βιομάζας, στηρίζονται σε μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο και αυτά περιληφθήκαν και στι ε, προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συνεργασία μεταξύ των ομάδων εργασία είναι πολύ σημαντική και λαμβάνει η χώρα και το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποδεικνύεται και εμπράκτως με την ε, οργάνωση αυτή τη δημόσια ακρόαση. Βέβαια κάποιε βελτιώσει ε, γίνονται και μπορούν να γίνουν. Ε, ένα από τα θέματα είναι ο κανονισμός για το LULUCF, χρήση γης, αλλαγή χρήσης γης και δασοκομεία. Δεν θα μιλήσω ε, λεπτομεριακά, πάντως έχουμε κάποιες απορίες για τις ε, πληροφορίες που στις οποίες στηρίχθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η βάση πληροφοριών ήταν κάπως ε, αβέβαιη και η κοινωνικο-οικονομική ανάλυση των επιπτώσεων ατελής. Υπάρχει λοιπόν κάποιο ζήτημα συνοχής ε, και αυτής της, ε, της νομοθετικής πράξης και τη υλοποίηση των στόχων κλίματος, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, απασχόλησης και ούτω καθεξής. Επίσης, μια αναλυτική μελέτη των επιπτώσεων των ευρωπαϊκών πολιτικών και της νομοθεσίας που επηρεάζουν τη δασοκομεία έγινε, αλλά δεν υπήρξε συνέχιση, follow-up. Το θέμα είναι, αν θέλουμε αποτελεσματικές πολιτικές, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη βάση πληροφοριών που θα στηρίζει αυτές τις πολιτικές. Και πού θα δώσουμε την έμφαση στο μέλλον, κατά τη γνώμη μας. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να ε, επικαιροποιήσουμε, να αναβαθμίσουμε το το συντονισμό και τη συνοχή των επόμενων πολιτικών και να συνεχίσουμε να αποδίδουμε ιδιαίτερο ρόλο στην ε, δασοκομεία σε ό,τι αφορά τη στρατηγική βιοοικονομία, στην αγροτική ανάπτυξη, την καινοτομία, τι επενδύσει κ.ο.κ. Επίση, να ενισχύσουμε την ε, βάση πληροφοριών, ένα ζήτημα ιδιαίτερα ευαίσθητο στα κράτη-μέλη. Αλλά πιστεύουμε ότι με βάση αυτή την ε, τομεακή προσέγγιση μπορούμε να βελτιώσουμε τη βάση πληροφοριών μα. Και επίση, να χρησιμοποιήσουμε πιο προηγμένες τεχνολογίες για να αναβαθμίσουμε αυτή τη βάση των πληροφοριών. Και θέλουμε η βιώσιμη ε, στρατηγική για τα δάση να δράζεται σε μια βιώσιμη πολιτική που θα, θα καλύπτει το σύνολο της αλυσίδας αξίας και θα εμπλέκει όλους τους φορείς σε τοπικό, εθνικό και ευρύτερο επίπεδο. Και τώρα θα πρέπει να αποφύγουμε την αποψήλωση και αντί να, να επικεντρωνόμαστε μόνο στα προβλήματα, να υιοθετήσουμε μια πιο θετική προσέγγιση και ένα σχέδιο δράσης για μια βιώσιμη δασική διαχείριση. Το βασικό ζήτημα είναι πώς θα ε, βελτιώσουμε στο μέλλον την εφαρμογή της ε, δασικής πολιτικής. Θέλουμε περισσότερες συνεδριάσεις της μόνιμης ε, δασικής επιτροπής, πιο εντατικό έργο και πιο καλή εφαρμογή αλλά καλύτερη και καλύτερη προετοιμασία. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνοχή και τη συνεργασία. Και γι' αυτό και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους ε, και να βελτιώσουν τις προσπάθειές τους. Και δεν θα πρέπει να τα αφήνουμε όλα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τα πραγματοποιεί σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να έχουμε και κάποια εγχειρήματα σε διεθνές επίπεδο και να αξιοποιήσουμε όλες τις διαθέσιμες διαδικασίες. Και τέλος, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Εμείς ε, προτείνουμε να συνεχιστεί η κοινή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Δασικής Στρατηγικής, να γίνει κατάλληλη αξιολόγηση τώρα και ελπίζουμε η στρατηγική για τα δάση να αποτελέσει σημαντική προτεραιότητα και στα μελλοντικά προγράμματα του Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίση θα πρέπει να συνεχίσουμε την έντονη προσπάθεια και στα υπόλοιπα φόρα, προκειμένου να αναδείξουμε τη σημασία των δασών σε όλε τι επιμέρου πολιτικέ. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στη συζήτηση. Το λόγο πρώτα ζήτησε ο κύριος Άγνιου. Παρακαλώ, ο κύριος Άγνιου. Ένα λεπτό παρακαλώ καθένας. Χαίρομαι που είμαι ο πρώτος ομιλητής, γιατί μάλλον ξέρετε τι θα πω. Θα πω ότι η δασοκομεία δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, δεν είναι κοινοτική αρμοδιότητα. Ακούγοντας όμως τις παρουσιάσεις αυτές, ο απλός πολίτης θα ε, θεωρήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τι ίδιες αρμοδιότητε για τη δοσοκομεία με αυτέ που έχει για τη γεωργία. Δεν ισχύει όμω αυτό. Και οι ευρωβουλευτέ που υποτίθεται ότι προσωπούν τους ε, ψηφοφόρου είστε συνένοχοι σε αυτή την παραπλάνηση που ε, επιχειρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχουμε δικαίωμα να συζητάμε τέτοια πράγματα. Δεν είναι κοινοτική αρμοδιότητα. Και αν το συνεχίσουμε θα δημιουργούμε προηγούμενο. Γιατί αν μπορεί να εμπλακεί σε αυτά και να παρέμβει σε θέματα δασοκομείας, γιατί να μην παρεμβαίνει και σε θέματα φορολογία, σχολικού προγράμματος, ε, ή στα, εθνικά συστήματα υγείας αν τις επιτρέψουμε τέτοιες παρεμβάσεις. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Το να ισχυριζόμαστε ότι θα βελτιώσουμε το παγκόσμιο κλίμα δεν είναι αρκετό επιχείρημα. Ε, εκτός και αν έχουν πάρει στραβό δρόμο τα κράτη-μέλη. Αλλιώς ε, θα πρέπει να αγνοήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για ασφαιδερισμό αρμοδιοτήτων. Ευχαριστώ. Ναι, όλοι το γνωρίζουμε. Αλλά κάποια θέματα συντονισμού και κάποια συνεργασία χρειάζεται για να βελτιώσουμε τη γενικότερη κατάσταση. Βάιτς. Σε αυτό το θέμα θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να νοιαστεί για τη δοσοκομεία, γιατί αν θέλουμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα του κλίματος θα πρέπει να εξηγήσω ότι επηρεάζουν και τα δάση. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο πρέπει να απασχοληθεί με αυτό το ερώτημα, να ασχοληθεί το ερώτημα. Και ένα άλλο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι δείχνουμε με το δάχτυλο μη ευρωπαϊκές χώρες όπου αποψηλώνουν ε, τροπικά δάση. Έχουμε όμως και εμείς τέτοιες περιπτώσεις στη Ρουμανία, στην Πολωνία και στην Ουγγαρία συμβαίνουν τέτοια πράγματα και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε πώς θα μπορέσουμε να ε, εφαρμόσουμε μια βιώσιμη διαχείριση. Πρέπει να προσπαθήσουμε στο μέλλον υπάρχει εμπλοκή και από τους περιβαλλοντολόγους και γι' αυτό θέλω να ευχαριστώ την Επιτροπή για, την χρήσιμη για το χρήσιμο έργο της. Ευχαριστώ. Μην ξεχνάτε ότι έπονται άλλε δύο ε, θεματικές ενότητες, ε, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Κύριο κύριος Φλάναγκαν. Ευχαριστώ πολύ για τον κύριο Παλάχη μια ερώτηση. Αναφέρθηκε σε μια αποτελεσματική επιστημονική πολιτική. Χαίρομαι που το είπε, γιατί και εγώ ήμουν υπέρμαχος της βιομάσας στη χώρα μου για τη δημιουργία ενέργειας. Από τότε έμαθα κάποια πράγματα ιδιαίτερα από τον καθηγητή της Έμψικεν από το Πρινστόν. είπε ότι και είναι βιομάζα στο Νιου και φαίνεται τελικά ότι δημιουργεί 70% περισσότερες εκπομπές του άνθρακα από ότι ο άνθρακας ο ίδιος. Και ο κ. Σέτσιγκερ αναρωτήθηκε μήπως θα έπρεπε να επιστρέψουμε στην καύση του άνθρακα. Απλά και μόνο. Και είπε ναι. Αν δείτε λοιπόν τα δεδομένα Ισχύει αυτό. Αλλά αν αρχίσει να το διαδίδει αυτό, το οποίο είναι αλήθεια, δεν θα μείνει στη δουλειά του και πολύ. Και το ίδιο ισχύει και με τα δέντρα, με την καύση των καυσόξυλων. Να ρωτήσω λοιπόν, τι σκεφτόμαστε να κάνουμε. Ακούσαμε, μάλλον θεωρούμε ότι ένα εκτάριο φωτοβολταϊκών θα δημιουργήσει ε, την ίδια ενέργεια με 100 εκτάρια ε, προϊόντος δασοκομείας. Α, το κινητό αυτό ήταν κόρη μου, έτσι. Ε, το λεπτό σας, κύριε Φλάναγκαν. Κυρία Μίλλερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα δασική θετική έχει ένα πρόγραμμα περιορισμένου χρόνου για τη βιώσιμη διαχείριση και για την περαιτέρω εξελίξη στον τομέα των, της καινοτομίας. Φυσικά η βιοπικιλότητα και η κλιματολογική αλλαγή είναι ένα σημαντικό τομέα, όμως θα πρέπει να δούμε και την ιδιοκτησία, το, να προσθέσουμε τους ιδιοκτήτε διασών, δασών γιατί έχουν μικρή επιρροή στις γενικές διευθύνσεις. Υπάρχει συνοχή. Και τα δικαιώματα των ε, ιδιωτών ε, λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της ε, διαλόγου για την κοινωνική ε, πολιτική της αλλαγής χρήσης γης και οι εμπειρογνώμονες εργάζονται εντατικά για να εκπροσωπήσουν ε, τους, ε, τους ε, του κλάδου. Ευχαριστώ κυρία Βιρκούνεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους καλεσμένους μας, τους εμπειρογνώμονες. Φυσικά ξέρουμε ότι η δασική πολιτική εμπίπτει σε εθνικές αρμοδιότητες, αλλά μια και ασχολούμαστε με νομοθετικές προτάσεις που αφορούν το κλίμα και το περιβάλλον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα δάση, που είναι σημαντικό το τμήμα της πολιτικής κλίματος και περιβάλλοντος. Μας είπατε ότι η δασική στρατηγική μας σε γενικές γραμμές είναι καλή. Ε, Ποιε είναι οι αδυναμίες, λοιπόν, κάποια στοιχεία από τη στρατηγική μας για τα δάση που θα μπορούσαμε να τα προσθέσουμε και να την εμπλουτίσουμε. Επίσης, μας είπατε ότι ακόμη και αν το βασικό στοιχείο είναι ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη συνοχή και καλύτερο συντονισμό με την, στρατηγική, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δάση, ίσως παρά είναι αδύναμη, δηλαδή δεν επηρεάζει επαρκώς τις πολιτικές μας και την προετοιμασία, τη χάραξη των πολιτικών, όπως θα έπρεπε περισσότερο. Επίσης είπατε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρογνωμοσύνη της μόνιμης ε, Επιτροπής για τα δάση κατά την ε, προετοιμασία των πολιτικών και τη μελέτη των επιπτώσεων. Έχετε άλλες συμβουλές για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις μελέτες αντικτύπου που κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να λαμβάνουν υπόψη και τον αντίκτυπο στα δάση. Κάποιο εμπειρογνωμονα είπε ότι η χρήση αλλαγή χρήση γη και η δοσοκομεία δεν ήταν καλό παράδειγμα γιατί η βάση πληροφοριών δεν ήταν άρτια. Έχουμε κάποια καλά παραδείγματα που ελήφθη υπόψη η εμπειρογνωμοσύνη τη μόνιμη δασική επιτροπή και έγιναν σωστέ μελέτε επιπτώσεων ώστε να λαμβάνεται υπόψη και ο δασικό κλάδο. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Παρακαλώ ε, ένα λεπτό, το πολύ ενάμιση, αλλά όχι παραπάνω. Κύριος Αντριέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σα ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία και τους δύο πρώτους εισηγητές. Καταρχάς, επειδή έστω και δεν είναι άμεση αρμοδιότητά μας, είναι και η κληρονομιά. Το πήγε η Κομισιόν ότι τα δάση είναι δόση για το περιβάλλον και για την κλιματική αλλαγή. Να το πενθυμίσουμε αυτό και νομίζω είναι κέριο να πούμε ότι οι προσανατολισμοί που βάλαμε το 2015 για την πολιτική των δασών της Ένωσης πρέπει να αξιολογηθεί πιο ισχυρά, πιο έντονα. Επίσης θα πρέπει να έχουμε κριτήρια βιωσιμότητας για τα δάση στην Ευρώπη. Πρέπει να δούμε και τι γίνεται και να δούμε επίσης και τα φόρουμ τα ευρωπαϊκά που χρησιμοποιούμε να λειτουργούν σωστά. Live, FSR και άλλα προγράμματα και η χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων ακριβώς πώς αξιοποιείται στα πλαίσια των δασών. Ευχαριστώ. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι ανανεώσιμα τα δάση, αλλά πρέπει να δούμε το σύνολο του κύκλου και υπάρχουν πολλές μελέτες που έχουν γίνει σχετικά, αλλά λέμε ότι έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Ενέθε λοιπόν ότι η πολλαπλή χρήση του, της ξυλίας και του δάσους ε, είναι αντικείμενο αυτών των μελετών, αλλά νομίζω ότι σήμερα πια πρέπει να πάμε παραπέρα. Δηλαδή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έστω και είναι εθνική αρμοδιότητα, και αντίθετα με τους προαλήσατες, θεωρώ ότι η Ευρώπη θα πρέπει, το είπε ο κ. δεν είναι αρμοδιότητα, αλλά εμείς θα πρέπει να αναλαμβάνουμε αυτή την αρμοδιότητα. Και θα πρέπει να δούμε σήμερα πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της χρήσης ε, της γης ή μέσω άλλων δράσεων, ο Επίτρος κλπ. θα μπορούσαν να παρανεύουν σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Και τώρα η κυρία Ματίνα Κοβέρκα ε, είναι πρόεδρος της ομάδας εργασίας ε, της ΚΟΠΑ ΚΟΖΕΚΑ για τη δασοκομεία. Παρακαλώ, ο κύριος μάλλον, συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω μια μικρή δήλωση. Διαπιστώνω ότι θα κάνουμε λόγο για την κλιματική αλλαγή, κάνουμε λόγο για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων, αντί να συζητήσουμε πώς θα διαμορφώσουμε το ενεργειακό μέλλον στην Ευρώπη και πώς θα πρέπει να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο η δασική πολιτική. Η ανησυχία μας είναι ότι αυτά που συζητώνται σε άλλους τομείς σε σχέση με τα δάση θα πρέπει να είναι σχετικά και συμβατά, να μην υπάρχουν αντιφάσεις και να, θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ιδιοκτήτες ε, δασών, τους δασοπόνους, να τους ενισχύσουμε ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Έχουμε ένα, μια πολυλειτουργική δασική οικονομία η ισχύ της Ευρώπης στους πόρους είναι τα δάση και είναι κάτι που θα πρέπει να αποδυναμώσουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν επιγόντως μια στρατηγική γιατί χρειαζόμαστε την βιοενέργεια, ε, ε με, ε, από τα δάση. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Και πάλι θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ε, διακεκριμένους μας εμπειρογνώμονες για να απαντήσουν. Με όποια σειρά θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις Ξεκινώ από το θέμα της βιοενέργειας των δασών. Για το θέμα αυτό της βιοενέργειας από τα δάση θα χρειαζόμαστε ολόκληρη μέρα για, να, για συζήτηση, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο και είναι πολύ διαφορετικά πράγματα που εντάσσονται σε αυτή την έννοια. Τη βιοενέργεια από τα δάση. Δεν μπορούμε να, να πούμε μονοσήματα αν είναι καλή ή κακή. Και σε μερικές περιπτώσει ε, θα έχει νόημα. Σε πολλές ε, περιπτώσεις άλλε δεν θα έχει νόημα. Όπως είπα όμω και προηγουμένω στην ομιλία μου, μακροπρόθεσμα ε, ο συγκεκριμένος πόλος για το δασικό τομέα είναι να αντικαταστήσει υλικά όπως το τσιμέντο, χάλιβας ή άλλα που στηρίζονται στον άνθρακα υλικά ανανεώσιμα, όπως το ξύλο. Τώρα, ε, στις ε, συζητήσεις ε, δεν είναι ένα θέμα που πρέπει άπαξ να διαθετηθεί. Χρειαζόμαστε ένα συνεχή διάλογο. Πολλό δε μάλλον που οι προσδοκίες για τους πόρους του δάσους αυξάνονται. Και είναι όλο και περίπλοκο το περιβάλλον της πολιτικής, αλλά υπάρχει και αύξηση της παραπληροφόρησης. Και σε αυτό το διάλογο πολιτικής ε, θέλουμε μια διορατική και προορατική προσέγγιση. Θα πρέπει γι' αυτό να έχουμε έναν επιστημονικό διάλογο έντιμο ώστε να ενημερώνονται οι, πολιτικοί θύναντες. Και αυτό λείπει στην δασική στρατηγική και στις υπάρχουσες ε, κυβερνητικές δομές. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της δασικής στρατηγικής, όπως είπα, το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Δάση είναι αξιόλογο, έχει πολλά εύστοχα σημεία, αλλά το βασικό ερώτημα είναι, είναι ε, στρατηγικό σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της δασικής πολιτικής στην Ευρώπη. Ε, ο συνάδελφος αναφέρθηκε σε κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναλήφθησαν. Ίσως όμως δεν εξετάστηκε, ε, δεν εξετάστηκε σαφές δεόντως η στρατηγική πολιτική. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα δασοκομεία στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη τη Υπέθρου, πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ είναι διαθέσιμα, με 5% των συνολικών δαπανών, 5% λοιπόν ε, του προγράμματος καλύπτει το 40% της επικράτειας του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Επίσης, αυτά τα 7 δισεκατομμύρια, τι επιπτώσεις έχουν στην Ευρωπαϊκή Δασική Στρατηγική. Θα πρέπει να γίνει μία ε, ε, δελεχής ανάλυση, κάτι που ξεκίνησε, για να δούμε πόσο αποτελεσματικά είναι τα μέτρα της δασοπονίας που εφαρμόζουμε. Αυτά από μένα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Ένα σημαντικό ζήτημα πολιτικής είναι το θέμα της αρμοδιότητας. Αλλά στο αφήσουμε προς το παρόν, γιατί εγώ θα σχολίζα το εξής. Έχουμε διάφορες πολιτικές που ασχολούνται με θέματα νοσοκομείας και το πώς χαράχτηκε η αντίστοιχη ευρωπαϊκή στρατηγική. Σας καλώ λοιπόν όλους να διαβάσετε Κάτι που με πολύ ωραίο τρόπο το περιγράφει σε μια σελίδα. Δηλαδή για το πώς και γιατί χρειάζεται, γιατί χρειάζεται όλο αυτό το πλαίσιο. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, δεν συγκράτησα τα ονόματά σας, να προσπαθήσω όμως να απαντήσω. Νομίζω ότι υπήρξε μια ερώτηση για τα θετικά και για τα κενά της στρατηγικής της Ένωσης για την δασοκομεία. Η στρατηγική αυτή δεν είναι ένα απλό έγγραφο το οποίο βγαίνει και μπαίνει μετά στο αρχείο. Έχει στόχους που πρέπει να εφαρμοστούν. Τώρα, κατά πόσο αυτοί οι στόχοι εφαρμόζονται, θα πρέπει να το δούμε σε συνάρτηση των εξελίξεων και των προσαρμογών που πρέπει να κάνουμε. Οπότε εδώ θα πρέπει να δούμε τη οικονομική στρατηγική πούμε, για τα δάση όταν εξετάζουμε το πλαίσιο της ανάπτυξης της υπαίθρου ή όταν συζητάμε για προγράμματα βιοπικιλότητας. Εκεί ακριβώς θα πρέπει να ενσωματώσουμε την προοπτική, την συνιστόσα, την πτυχή της δασοκομείας. Επίσης υπήρξε το ερώτημα του κατά πόσο Έχουμε καλά παραδείγματα όπου μπόρεσε η Επιτροπή Δασοκομείας να ασκήσει επιρροή. Αναφέρθηκα σε μια ομάδα εργασίας εγώ προηγουμένως που ασχολήθηκε με το θέμα και τα κριτήρια που υπάρχουν εκεί της βιωσιμότητας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με αυτή την προσέγγιση και αυτό είχε περιληφθεί στην πρόταση της ε, Κομισιόν για τη βιομάζα και την ενέργεια. Επίσης υπάρχουν θετικές εμπειρίες μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος ε, ε, Πληροφόρησης για τα δάση. Αυτό δεν αφορά μόνο τη χώρα μου, αλλά έχουμε πολλές θετικές εξελίξεις και αλλού. Θεωρούμε λοιπόν ότι και αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας. Επίσης, για τα βιώσιμα κριτήρια και την χρήση του στο παρελθόν στα πλαίσια της πολιτικής για τα δάση στην Ευρώπη. Για τα κριτήρια. Νομίζω ότι αυτά εφαρμόζονται και ελπίζω με αυτά που είπα τώρα να απάντησα τουλάχιστον σε κάποιε ερωτήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά τους εμπειρογνώμονες μας για τις παρουσιάσεις τους και ευχαριστώ και τους συναδέλφους ε, για τις ερωτήσεις. Περνάμε στο δεύτερο τμήμα, στο οποίο θα προεδρεύσει η κυρία Κούμπουλα Νάτρη από την ε, Επιτροπή Ήτρε. Παρακαλώ. Έχουμε μείνει πέντε λεπτά πίσω σχέση με το χρονοδιάγραμμα εκ μέρους του κυρίου Μπούζεκ, του Πρόεδρου της Επιτροπή Ήτρε, που κολλείεται. Θα ήθελα, θα να σας πω πόσο εκτιμούμε αυτή την συνδιοργάνωση της ε, δημόσιας ακρόασης με θέμα την Ευρωπαϊκή Δασική Στρατηγική που γίνεται για δεύτερη φορά. Το εκτιμούμε ιδιαίτερος. Στο δεύτερο τμήμα θα μιλήσουμε για τον δασικό κλάδο στη βιοοικονομία, τις μεταπητικές βιομηχανίες και την καινοτομία. Δύο είναι οι ομιλητές μας στο τμήμα αυτό. Έχουμε πρώτα τον κύριο Γκούτεμπερκ που είναι πρόεδρος των Γερμανών Ιδιοκτήτων Δασών και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ιδιοκτήτων Δασών ασχολείται με τη διαχείριση του δάσου, ε, την οικολογία και έχει σπουδάσει η φιλοσοφία της οικονομίας. Παρακαλώ κύριε Γκούτεμπερκ, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Αρχικά θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για αυτή τη διασυσμική πρωτοβουλία να έχετε αυτή την κοινή ακρόση σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι η Δεύτερον, σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσετε ως εκπρόσωπο των ιδιωτικών ιδιωτικών δασών για να σας μιλήσω για τις δικές μας προσδοκίες και τα οράματα τα οποία, τα μεγάλα οράματα όπως ξέρουμε είναι απλά ποιοι είμαστε εμείς, ποιοι είναι οι ιδιότητες, ιδιότητες διασών. Δεν γινόμαστε και πολύ αντιληπτοί. Αν και είμαστε πολλοί, είμαστε 16 εκατομμύρια άτομα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλο νούμερο, αλλά ε, μικροϊδιοκτήτες. Το μέγιστο μέγεθος, το κατά μέσο όρο μέγεθος ε, ιδιοκτησιών ανέρχεται σε 5 με 6 γήπεδα ποδοσφαίρου και γι' αυτό είναι και μεγάλες οι προκλήσεις. Η μεγάλη πυκλομορφία στους προσωπικούς στόχους που έχουμε για το τι θα κάνουμε τα δάση μας. Παρ' αυτά είμαστε ενωμένοι, σεβόμαστε τις ε, φυσικές διαδικασίες που βιώνουμε καθημερινά στα δάση μας και υπάρχει ένα πράγμα που έχουμε μάθει ε, στο πέρασμα των γενεών, ένα πράγμα που υπερισχύει κάθε εικονική ιδεολογίας. Η βιώσιμη διαχείριση διασών είναι εφικτή μόνο αν την προσεγγίσουμε με έναν πραγματικά ολιστικό τρόπο. και να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα θέματα. Όταν κάνουμε λόγο για ολιστική προσέγγιση, ε, εννοούμε ότι πρέπει να βρούμε μια ισορροπία, μια μέση λύση, μια χρυσή τομή. Η μεγιστοποίηση ενό των τριών πυλώνων αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε κατάρρευση του συστήματο. Τα δάση μα είναι από τα πιο ταλαντούχα οικοσυστήματα. Παράγουν οξυγόνο, συλλέγουν νερό, καθαρίζουν, σταθεροποιούν το ε, έδαφος, φιλοξενούν ε, χλωρίδα και πανίδα, είναι αρχιτέκτονες ε, τοπίου και είναι κέντρα αναψυχής και εκπαίδευσης και φυσικά ε, μας δίνουν ένα από του σημαντικότερους ανανεώσιμους πόρους, το ξύλο. Έχει υποθεί ότι ο 21 ο αιώνας θα είναι ο του ξύλου και συμφωνώ απόλυτα με αυτό το όρομο, μόνο αν μπορούμε να συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε τα δάση μας και να μην ακολουθούμε κοντόφθαλμες ε, τάσεις της εποχής. Ως ιδιοκτήτες επενδύουμε χρήματα σε δέντρα τα οποία χρειάζονται 100 χρόνια για να μεγαλώσουν. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι χαζό. Αλλά οι πολιτικές που αλλάζουν κάθε 5 με 10 χρόνια δεν βοηθούν στην πραγματικότητα, ούτε μας κινητοποιούν για να το συνεχίσουμε αυτό και στο μέλλον. Τα τελευταία 300 χρόνια σταδιακά βελτιώσαμε τις γνώσεις μας ε, για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, Βέβαια, εξακολουθούμε να μαθαίνουμε σε καθημερινή βάση, αλλά παράλληλα έχουμε δώσει αρκετά πιστήρια ότι μπορούμε να παράγουμε ξύλο χωρίς να επηρεάζουμε αρνητικά ε, άλλες δραστηριότητε των δασών. Επίσης είμαστε πολύ ανοιχτοί στις πρακτικές ε, συμβουλές από ενδιαφέρομενα τρίτα μέρη που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας και, ε, και, τα δάση. Ωστόσο, αυτό που δεν μπορούμε να ανεχτούμε και δεν εκτιμούμε είναι οι εκ των υστέρων απαιτήσει, καθοδηγούμενε από ιδεολογίε και όχι από επιστημονικά δεδομένα και εμπειρική γνώση. Ω ιδιοκτήτε δασών, έχουμε την ευθύνη για το περιβάλλον μα και επίση φέρουμε και τον οικονομικό κίνδυνο. Αυτή είναι η διαφορά, η βασική, ανάμεσα σε εμά και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη και γι' αυτό ζητάμε μια προτιμησιακή ε, προσέγγιση σε σχέση με τα δικαιώματά μας. Το 1996 και μάλιστα ένα μέλος ε, αυτού του κοινοβουλίου, ο Σέρ Ντέιβιντ Τόμας, ο οποίος τόνισε στην έκθεσή του στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο ότι η τη της τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονό ότι τα περισσότερα δάση τη Ευρώπη είναι η διεκτησία εκατομμυρίων διοκτητών δασών που πρέπει να ε, εξασφαλίσουν μια πολυλειτουργική διαχείριση των δασών και την βιωσιμότητα των σχετικών ε, πόρων. Αυτή η διοκτήτης λοιπόν πρέπει να είναι σεβαστή. Σήμερα οι συστάσεις του εξακολουθούν να είναι επίκαιρες. Η πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική, δασική στρατηγική, έδωσε ένα ξεκάθαρο σήμα να γίνει σεβαστός ολιστικός χαρακτήρας της ε, δοσοκομείας και να λάβει υπόψη την αρχή της επικουρικότητας. Αυτά τα δύο σημαντικά θέματα σήμερα είναι δευτερεύουσα σημασίας στην τρέχουσα πολιτική για τα δάση, καθώς τα δάση και τα σοπονία φαίνεται ότι εξυπηρετούν άλλους τομείς της πολιτικής. Και αυτό φαίνεται στις καθημερινές διαβουλεύσει που γίνονται στο πλαίσιο του Λούλου, ΣΥΕΦ, του ΡΕΔ 2 και άλλων πολιτικών. Είμαστε επιπισμένοι ότι η Ευρωπαϊκή Δασική Πολιτική μπορεί και θα μπορούσε να ε, οδηγήσει μια πιο ισορροπημένη πολιτική. Αν τη λάβουμε σοβαρά υπόψη, συνοχή. Αυτό ήταν ο βασικός τη στόχος και προφανείς δεσμοί ε, της Αντικής με τους στόχους εφόρους ανάπτυξης του ΟΗΕ και της Συμφωνίας του Παρισιού είναι πολύ σημαντικά για τον συνεχή σχεδιασμό της ευρωπαϊκής πολιτικής ασχέτου του τομέα. Επίσης, η αναθεώρηση της ε, ε στρατηγικής τη βιοοικονομία θα μπορούσε να υποστηρίξει την ολιστική προσέγγιση της ε, δασικής στρατηγικής. Είναι στο χέρι μας με τα καταναλωτικά, τις καταναλωτικές μας συνήθειες να συνεχίσουμε να έχουμε αρνητικές επιπτώσεις. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στους φυσικούς πόρους ε, που μπορούμε να διατηρήσουμε βιώσιμα στο, στο χώρο μας. Η βιωσιμότητα δεν μπορεί να ανατεθεί στο εξωτερικό. Τα δάση είναι κομμάτι της υπαίθρου και είναι η βασική πηγή ανάπτυξης και παραγωγής υλικών και προϊόντων σε μια μεγάλη ποικιλία παραδοσιακών ε, και καινοτόμων ε, ε, ληστών αξίας. Και οι πρόγραμμα μας επένδυσαν πολύ σε, στα δάση για οικοδομικά υλικά και για άλλα προϊόντα τα ίδια δάση κοιτάμε κι εμείς αρκετές γενναίες μετά για να παρέχουμε επίσης δομικά υλικά, βιοενέργεια, προϊόντα υγιεινής, ε, ε υλικά υψηλής τεχνολογίες, ίνες για την υφαντουργία, για να ονομάσουμε, το ονομάσουμε κάποια από αυτά. Είναι μία έξυπνη, ένα έξυπνος πόρος στα δάση και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ε, μια πολύ ισχυρή στρατηγική που θα συμπεριλάβει όλου αυτού του πολύπλοκου τομεί πολιτική. Νομίζω ότι στην Ευρώπη ξέρουμε πώ να διαχειριστούμε με βιώσιμο τρόπο τα δάση μα και στον 21ο αιώνα θεωρώ ότι το οφείλουμε στι επόμενε γενιέ να παρέχουμε το σωστό συνεκτικό πλαίσιο και να ε, αναδείξουμε το ξύλο και τα δάση σε έναν από του πιο, ε, πιο σημαντικούς ε, πόρους. Ευχαριστώ πολύ. <laughs> Σε έμεινα και 30 δευτερόλεπτα. Ο επόμενο είναι ο κύριος Κόρα Τομασεύσκη. Επίσης έχει δοκτορά σε, στην επιστήμη των δασών, γιατί μιλούμε για επιστήμη και είναι και σύμβουλος του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας στην Πολωνία και γενικό διευθυντής του Εθνικού Οργανισμού Διαχείρισης Κρατικών Δασών της Πολωνίας. Πάνω από 40 χρόνια δραστηριοποιείται στο στο δασικό τομέα. Παρακαλώ κύριε και έχετε το λόγο. Ε, ε, ευχαριστώ. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, αντίθετα με τον προλαλήσαντα, εγώ εκπροσωπώ μια διαφορετική κατάσταση. Δηλαδή, σε εμά ε, η κυρίαρχη μορφή ιδιοκτησία είναι η κρατική ιδιοκτησία των δασών. Στην Πολωνία δηλαδή έχουμε περίπου 90 εκατομμύρια εκτάρια δάσους. Ε, τα περισσότερα, η συντηρητική πλειοψηφία είναι κρατικά δάση και μόνο 19% είναι ιδιωτικά δάση. Δηλαδή πάνω από 80% των ε, πολωνικών δασών είναι δημόσια δάση κρατικής ιδιοκτησίας. Εγώ συμφωνώ με πολλά από αυτά που αναφέρατε. Δηλαδή ότι η νέα δασική στρατηγική είναι μία ε, δράση ε, εκτελεστική, αλλά δεν έχει δεσμευτική αξία λόγω της μία έλλειψης ε, κοινοτικής αρμοδιότητας. Πάντως και ως μία αρμοδιότητα έχει κάποια αξία αυτή η επέμβαση. Όταν ε, διάβασα για πρώτη φορά την ε, νέα την ευρωπαϊκή στρατηγική, έμεινα ικανοποιημένο ω ε, διευθυντή του Εθνικού Οργανισμού Διαχείριση Κρατικών Δασών, γιατί θεωρώ ότι αυτή η ευρωπαϊκή στρατηγική συνάδει πλήρω με το πολωνικό δίκαιο για την δασική διαχείριση. Βέβαια, τις ε, παρούσες συνθήκες και τις πραγματικές και τις νομικές, αυτή η νέα δασική στρατηγική της ευρωπαϊκής στρατηγικής θα είναι πολύ δύσκολα πραγματοποιήσιμη ε, λόγω δύο παραγόντων. Καταρχήν, ε, λόγω κάποιων ε, αρμοδιοτήτων που εξακολουθούν να είναι κοινοτικέ και αφορούν κυρίως την πολιτική για το κλίμα, πολύ δύσκολο θα είναι να κρατήσουμε την έννοια της αηφόρου ε, δασικής διαχείρισης από το 2001. Γιατί μιλούμε για το τουλούλου ή αυτή, την χρήση γης, αλλαγή χρήση γης και δασοκομεία. Το επίπεδο όμως ε, ε, διαχείρισης των δασών και αξιοποίησης ε, της ξυλίας από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια τη ψηφοφορία και όχι με βάση τα δικαιώματα για τη φύση. Για παράδειγμα, στην Πολωνία θα πρέπει να μειωθεί ε, κατά ποσοστό η αξιοποίηση των δασών εξαιτία ακριβώ ε, ε, των κοινοτικών αρμοδιοτήτων. Και έτσι δεν θα στηρίζεται σε πραγματική γνώση τη διαχείριση ε, του δάσου και των αναγκών τη φύση, παρά σε συγκεκριμένη κατανομή μεταξύ ψήφων. Επίσης, η βιώσιμη δασική ε, διαχείριση ε, στην Πολωνία είναι παράδειγμα προς ε, μίμηση. Αν όμως δεν γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα της φύσης, αλλά περάσουμε σε διαχείριση με, μετά από ψηφοφορία, θα είναι πολύ δύσκολο να διαφυλάξουμε μια τέτοια βιώσιμη δασική διαχείριση στην Πολωνία. Επίσης, αν δεν παραμείνουμε σε αυτά τα όρια, θα μειώσουμε και το δικαίωμα της κατά το, την υπηρεσία της καταβόθρας διοξιδίου του άνθρακα που μέχρι στιγμής εξασφάλιζαν τα δάση και θα τα μετατρέψουμε σε παράγοντες που ενισχύουν τις εκπομπές άνθρακα. Θα πρέπει να προσέξουμε λοιπόν πώς εφαρμόζουμε τη νέα δασική στρατηγική. Υπάρχει ένας ε, οικολογικοκεντρικός ε, ε, παράγοντας, δηλαδή που τάσεται υπέρ μιας, ενός περιορισμού της παρέμβασης στα δάση με το επιχείρημα ότι η φύση αυτορυθμίζεται. Αυτό όμως δεν ισχύει γιατί μετά από κάποιες βιομηχανικές διαδικασίες αλλά και κάποιες διαδικασίες αστικοποίησης στα πλαίσια της ανάπτυξης του πολιτισμού είχαμε κατακαιρματισμό των δασικών μας περιοχών. Έτσι ε, έμειναν κάποιες νησίδες, περίπου 500.000 εκτάρια ε, στη βορειοκεντρική Ευρώπη έχουν μείνει ε, και μόνο ε, σε λίγα τέτοιες νησίδες έχουμε πραγματικά φυσικές διαδικασίες. Στα περισσότερα δάση δεν έχουμε ε, αρχαίγωνα δάση, στις περισσότερες περιοχές δεν έχουμε αρχαίγωνα δάση στην Ευρώπη, δηλαδή δάση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ελάχιστο είναι το δικό τους ποσοστό. Επίσης έχουμε κατακαιρματισμό της δασικής ε, διαχείρισης. Και μόνο με την ε, επέμβαση στη δασική διαχείριση μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη δασική πολιτική, όχι αφήνοντας τα δάση σε μια ελεύθερη ε, φυσική αυτορύθμιση. Επίσης θα πρέπει να ε, προστατεύσουμε και την περιβαλλοντική τους αξία αλλά και την κοινωνική αξία των δασών. Και αυτό το καταφέρουμε χάρη στις επεμβάσεις μας. Παρά λοιπόν κάποια αρνητικά σχόλια που ακούστηκαν στην Πολωνία, υλοποίησαμε αυτή την νέα ευρωπαϊκή δασική στρατηγική. Και θέλουμε στην COP24 να παρουσιάσουμε την δική μας ε, αντίληψη για την οικονομική πολιτική, οικονομική διαχείριση των δασών υπό το πρίσμα του άνθρακα. Και με κάποιες ε, επιπρόσθετες δραστηριότητες μπορούμε να ελοπίσουμε 31% του στόχου της μείωσης του διοξίδιου του άνθρακα. Και μάλιστα με προαιρετική εφαρμογή από το 2020, ε, ε, αποδεικνύοντας ότι η δική μας μέθοδος, η οικονομική μέθοδος διαχείρισης των δασών με βάση τον άνθρακα μπορεί να αποφέρει καρπούς και να μειώσει τις εκπομπές του άνθρακα στα επιθυμητά επίπεδα. Επίσης, ε, αυτή η αλυσίδα για ε, ξυλίας ε, και αλυσίδας αξίας στα πολωνικά δάση και την πρόθεση της χρήσης του ξύλου ως δομικού υλικού. μάλιστα, στο μέλλον θα αξιοποιούμε κυρίως αυτή την τεχνολογία της κατασκευής σπιτιών από ξύλο. Και μάλιστα υπάρχει ένα μεγάλη εμβέλεια σχέδιο για την πρόθεση αυτή του ξύλου υλικού στην Πολωνία. Επίσης έχουμε ε, την ενεργειακή λειτουργία ε, του ξύλου. Γιατί πολλοί μιλούν για το ενεργειακό ξύλο. Αλλά κανένας δεν θέλει να ε, καταλήξουμε σε ένα νομικό ορισμό του ενεργειακού ξύλου. Περιμένουμε εδώ και χρόνια αυτό τον ορισμό και μάλιστα τα κρατικά δάση της Πολωνίας ε, από το 1980 ε, αξιοποιούν ξύλο που κυρίως έχει ενεργειακό σκοπό χρησιμοποιώντας το ξύλο για την παραγωγή θερμότητας. Επίσης, έχουμε πολλές μορφές οργανωτικές και νομικές για την άσκηση της δασικής διαχείρισης. Αναφέρθηκε πριν από λίγο η, έκταση, μεγάλη έκταση των δασικών πυρκαγιών φέτος. Είχαμε πραγματικά μια φυσική καταστροφή στην Πολωνία. Χάσαμε 80.000 εκτάρια δασών από δασικές πυρκαγιές. Και είναι 1,5% η έκταση της Βαρσοβίας. Είναι πραγματικά ήταν μεγάλη καταστροφή και παρόλα αυτά, χάρη στην σωστή και βιώσιμη ε, δασική διαχείριση που έχουμε στην Πολωνία, θα αντιμετωπίσουμε αυτή την φυσική καταστροφή. Και παρόλα αυτά, ε, θα χάρη στην πολιτική μας θα μετατρέψουμε σε, τοπία, ε, σε πάρκα τοπίου αυτά τα πάρκα φυσικής καταστροφής που δημιουργήθηκαν μετά τις ε, δασικές πυρκαγιές. Ευχαριστώ. Όπως σας είπα, 8 λεπτά έχει ο κάθε ομιλητής στη διάθεσή του. Παρακαλώ να το σέβεστε αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτή ήταν η δεύτερη φάση της ακρόασης. Ε, ο κύριε Σκοτ Κάτω. Ευχαριστώ. Μας δείξατε τις εικόνες των όμορφων δασών σας και κατάλαβα ότι εμείς αποψηλώσαμε τα δικά μας στη χώρα μου πριν πολύ καιρό και χαίρομαι τα δικά σας στην καλύτερη κατάσταση. Για τη συμβατότητα με τη συνθήκη του Παρισιού της πολιτικής για τα, δάση, για τα δάση. Οι ρυθμοί εξόριξης σε σχέση με τον αριθμό απορρόφησης δεξιδίου από τα δάση συμβαδίζουν και μιας και μιλάμε για στόχους διατήρησης της φύσης και βιοπικιλότητα για την Πολωνία. Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή καταλαβαίνω ότι το ποσοστό κάλυψης αυξάνεται στην, στην Πολωνία, όπως ε, ταυτόχρονα όμως μειώνονται και οι προστατευόμενες ε, περιοχές. Από τη στιγμή που έχουμε 9 εκατομμύρια εκτάρια, γιατί επιμένετε στο να υλοτομείτε μικρές περιοχές, οι οποίες είναι πολύ πλούσιες σε ε, βιοπικιλότητα και αποτελούν ευρωπαϊκή κληρονομιά. Και ε, οι πολιτικές εξόριξης έχουν επηρεαστεί καθόλου από το ημερήσιο πρόστιμο 100.000 ευρώ από το δικαστήριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση στην κυρία Γκούντεμπερικ, στον κύριο Γκούντεμπερικ. Αν υποστηρίζουν οι ιδιώτες διοκτήτες ε, την ε, τη συμφωνία την οποία την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν οι άλλοι τομείς πολιτικής επεμβαίνουν σε θέματα ιδιοκτησία. Κάνατε λόγο για ιδεολογία και υπερίθμιση Πιστεύετε ότι είναι παρικέ αν κάνουμε επιστημονικέ εκτιμήσει, τι σημαίνει βιώσιμη διαχείριση κτλ. Και μπορούμε να προσταθούμε από την υπερίθμιση ή θεωρείτε ότι δεν θα πρέπει οι άλλοι τομείς της πολιτικής να επεμβαίνουν στον τομέα της δασοκομείας. Ευχαριστώ κύριος Μπάιτς. Η ερώτησή μου απευθύνεται στον κύριο Ταματσίευσκη, Γενικό Πώς μπορείτε να μου εξηγείτε σε μια περιοχή προστατευόμενη του Νατούρα... γίνεται εξαπάτηση. Παρακαλώ, εξηγήστε. Ε, ο κύριο Κούσμιουκ. Εγώ έχω μια ερώτηση προ τον κύριο Τομασεύσκη, τον Διευθυντή του Πολωνικού Οργανισμού Διαχείριση Κρατικών Δασών. Στη Συμφωνία των Παρισίων αναφέρθηκε ο ρόλος των δασών ω παραγόντων μείωσης του διοξιδίου του άνθρακα. Κάτι τέτοιο δεν προβλέπει η ευρωπαϊκή δασική στρατηγική. Ε, τι γνώμη έχετε γι' αυτό. Ο κύριος Λίντς. Ευχαριστώ. Στον κύριο Κούτεμπεργκ μια ερώτηση. Καταστείτε σαφές Ε, για την πολυλειτουργικότητα του δάσους, κάνετε αναφορά στην αρχή της επικουρικότητας. Αυτό που καταλάβουμε είναι ότι υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις και προτάσεις νομοθετικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες παρεμβαίνουν στη δασοκομεία και αναφέρουμε στο ΛΟΥΣΙΕΦ τον τρίτο πυλώνα της κλιματικής πολιτικής. Κατά την άποψή σας, δεν να μου πείτε αν αυτή η πολυλειτουργικότητα θα μπορέσει να εξασφαλιστεί μετά από αυτά τα νομοθετικά μέτρα. Ή αν θα δοθεί έμφαση σε μία λειτουργία. Uh, Παρακαλώ, δυόμιση λεπτά έχετε οι δύο καλεσμένοι για να απαντήσετε για να ολοκληρώσουμε και αυτό το τμήμα. Ο κύριος Κούτεμπερκ. Ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Να ξεκινήσω με την τελευταία για την πολυλειτουργικότητα και την χρήση γης που ανέφερε ο κύριος Λίντς. Η απάντηση είναι όχι. Το μέλλον της πολυλειτουργικότητας δεν έχει αναγνωριστεί πλήρως. Αν παγώσουμε ή περιορίσουμε τη γεννητικότητα για την ξυλία, αυτό δεν λαμβάνει υπόψη του την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του δάσους ένα από τα κυριότερα δηλαδή ζητήματα για την ανάπτυξη της Πέθρου και όπως είπα προηγουμένως ένα από τα κυριότερα ζητήματα όταν εξετάζουμε το πώς το διαχειριστούμε τα δάση και τους ιδιοκτήτες τους, πώς να τους δώσουμε κίνητρα ώστε να αξιοποιήσουν το πιο, το πόρο, το πιο χρήσιμο πόρο στην Ευρώπη. Αφενός και αφετέρου, αν δούμε τα δάση, η συλλογή άνθρακα είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να το δούμε γενικότερα σε σχέση επίσης και με το θέμα της καταβόθρας εξωδίου άνθρακα και τι γίνεται με την ανταπόκριση των θεσμών, ας πούμε, για τα μέτρα περιορισμού των τρύπων. Και αυτό νομίζω ότι λείπει ακριβώς στις προτάσεις για την χρήση της γης. Η κυρία Μίλλερ ρώτησε κάτι σε σχέση με το Forest Europe, την ευρωπαϊκή πολιτική για τα δάση. Τη χρειαζόμαστε. Γιατί αποτελεί τη μόνη νομική αναφορά που έχουμε. Όταν μιλήσαμε για συνοχή προηγουμένως και κάποιος άλλος βουλευτής ρώτησε γιατί τα χρειαζόμαστε όλα αυτά. Εμείς στις ευρωπαϊκές πολιτικές έχουμε γύρω στα 400 εργαλεία που ασχολούνται έμεσα ή άμεσα με τα δάση. Αν λοιπόν δεν θεσπίσουμε μια νομική αραφορά, τότε νομίζω ότι μπορούμε να θεσπίσουμε στόχους ή να ασχοληθούμε με την στρατηγική των δασών, αν δεν υπάρχει αυτή η νομική αναφορά δηλαδή. Νομίζω ότι θα πρέπει να ισχύει πανευρωπαϊκά αυτό, γιατί θα πρέπει βεβαίως να ρυθμιστεί και σε επίπεδο χωρών ώστε να αντιμετωπίσουμε σωστά το θέμα της επικουρικότητας και να το υλοποιήσουμε σε επίπεδο νομικά ζημευτικών συμφωνιών. Αυτή είναι η σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο αυτών εργαλείων. Η κυρία Κάτω ρώτησε κάτι σε σχέση με την συμβασιμότητα σχετικά με συμφωνία του Παρισιού και το ρυθμό εξορίξεων. Έχουμε 60, με 60 70% αύξηση, οπότε έχουμε εδώ πολύ περιθώριο. Στη Γερμανία πάντως δεν κάνουμε παραπάνω εξορίξεις. Οπότε ακολουθούμε αυστηρά την αρχή της βιωσιμότητας. Παρ' όλα αυτά, για τα ποσοστά υλοτόμησης. Έτσι, γι' αυτά μιλάω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ και στο και παρακαλώ. Ε, ε, είμαι ευγνώμων ε, στον ε, κύριο που αναφέρθηκε στην, στο δάσος Πιαλοβέτσκα. Υπάρχει μεγάλη παρανόηση ως προς την υλοτόμηση σε αυτό το δάσος Μπιαγοβιέτσκα, το αρχαίγωνο δάσος, εξού και η εσφαρμένη εντύπωση που έχει δοθεί. Η... Το δάσος Μπιαγοβιέτσκα δεν είναι ε, πάρκο αρχαίγωνου τοπίου. Ε, εδώ και πολλά χρόνια όλοι οι δασικοί πόροι ε, είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης επέμβασης. Δεν είναι αρχαίγωνο ούτε αυτό το δάσος. Και μάλιστα από πριν από το Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε στοιχεία που δείχνουν πως η, γερμανική αεροπορία επηρέασε ε, και έχει στοιχεία για τις ε, ανθρώπινες επεμβάσεις. Σχεδόν όλα μας τα δάση είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης ε, δραστηριότητας. Και με, με βάση αυτή την ανθρώπινη επέμβαση έχουμε μια μοναδική βιοποικιλότητα και στην Πολωνία. Δεν έχουμε αρχαία χρονοδάσους, αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα ισορροπημένης και βιώσιμης δασικής διαχείρισης. Γι' αυτό και δημιουργήσαμε τέτοια μεγάλη βιοπικιλότητα στα δάση μας και συγκεκριμένα και σε αυτό το δάσος. Ε, άλλωστε η ξυλία είναι ένα πολύ φιλοπεριβαλλοντικό ε, μέσο και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Επαναλαμβάνω λοιπόν δεν είναι αρχαίγωνο δάσος το δάσος της Μπιαγοβιέτσκα. Ε, μιλήσατε για ένα φυσικό τοπίο. Τι θα πει φυσικό τοπίο. το δασικό φυσικό τομείο είναι ένα τοπίο στο οποίο γίνονται διαδικασίες αυτορύθμισης. Τέτοιες όμως διαδικασίες αυτορύθμισης που σας είπα θα γινόταν αν ε, είχαμε ε, στην Ευρώπη δάση ενός με δύο εκατομμυρίων εκταρίων. Αλλά ε, δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις πολλές στην Ευρώπη, γιατί έχουμε κατακαιρματισμό της δασικής διαχείρισης στην Ευρώπη και το δάσο Μπιαγοβέτσκα είναι μια νησίδα. Δεν έχουμε ε, τέτοια απομεινάρια αρχαίγωνων δασών. Αλλά απλώ εφαρμόστηκαν ε, διάφορες μέθοδοι δασικής ε, διαχείρισης. Τα κρατικά δάση και συγκεκριμένα το κρατικό δάσος της Μπιαγοβέτσκα δεν δέχεται διαδικασίες υλοτόμησης. Δεν γίνονται υλοτομήσεις εκεί, αλλά εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα εμ, δραστηριοτήτων προστασίας όπως προβλέπει η Natura 2000. Επειδή όμως είχαμε μεγάλα κρούσματα ε, κατά, ε, ε, αποψήλωσης λόγω της δράσης των σκαθαριών, τελικά είχαμε ε, τοπίο θεομηνίας στα κονοφόρα της Βιογοβιέσκα και δεν είχαμε τοπίο, πάρκο τοπίου. Δεν μπορείτε λοιπόν να μου λέτε ότι επίθεση από τα σκαθάρια αυτά που κατέφαγαν μεγάλο αριθμό του δάσους Μπιαγοβιέτσκα είναι αποτέλεσμα φυσικού τοπίου. Μάλιστα ε, θα παρουσιάσουμε την υπόθεση και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εμείς όχι μόνο δεν καταπατούμε ή δεν μειώνουμε τη βιοπικιλότητα, αλλά προσπαθούμε να την αποκαταστήσουμε γιατί εξαιτία της μεγάλης θεομηνίας ε, της φυσικής καταστροφής λόγω των σκαθαριών είχαμε μεγάλη επιδείνωση του τοπίου στο δάσος ε, Μπιαγοβιέσκα. Είχαμε μάλιστα 200 εκατομμύρια τέτοιες υλοτόμες. Ε, Αυτά δεν τα καταλαβαίνετε, λόγω των σκαθαριών. Σε καμία περίπτωση δεν εξαντλήθηκε βιοπικιλότητα και μάλιστα θα αποκαταστήσουμε τα οικοσυστήματα ε, και της χλωρίδας και της πανίδας ε, που ε, πλήγησαν. Δεν δεν πρόκειται που δεν είναι να καταστρέψουμε τη βιοπικιλότητα στο δάσος αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα την Συμφωνία των Παρισίων και την πολιτική Λουλουσιέφ, εμείς στην COP24 θα αποδείξουμε ότι η δασική διαχείριση και με βάση τον άνθρακα θα αποτελέσει τρόπο υλοποίησης των δεσμεύσεων του Παρισιού. Και θα δείξουμε πώς θα συμβάλλουν τα δάση στην, ε, στην αρέωση της συγκέντρωσης του διοξείδιου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο τρίτο τμήμα της ακρόσης, και θα, όπου θα περιδρεύσει ο κύριος Παύλ Πότς. Περνάμε στο τρίτο τμήμα της ακρόσης, λοιπόν. Θα επικεντρωθούμε στον περιβαλλοντικό ρόλο των δασών, στις υπηρεσίες οικοσυστήματος που προσφέρουν, στη βιοπικιλότητα και το καθεξής. Έχουμε δύο ε, εμπειρογνώμονες, την κυρία Χάνα Άχο, που είναι ακτιβίστρια για τα δάση και το κλίμα, και συμμετέχει στο δίκτυο ε, των δασών και των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουμε και την κυρία Γιάννα Μπέκ από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκη, ε, πρόεδρο της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για το Συμβούλιο Επιστημών. Είμαι εδώ για να μιλήσω για την κλιματική αλλαγή και τα δάση. θετικό μήνυμα είναι ότι τα δάση πράγματι έχουν τη δυναμική να μας, μας βοηθήσουν να μείνουμε κάτω από δύο βαθμούς. Όντω, αυτό το διάστημα τα δάση ε, τη Ευρώπη κατεβάζουν θερμοκρασία, αλλά τα δάση μπορούν παράλληλα να είναι αιτία υπερθέρμανση. Γιατί η αλλαγή χρήση ε, αφορούν το 40% της υπερθέρμανσης από το 1750 και αυτό συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν δούμε όμως τροπικά δάση, η διαχείριση των δασών έχει συμβάλει ε, επίσης ε, στην υπερθέρμανση και γι' αυτό έχουμε ε, μια αυξανόμενη δασική έκταση. Ο λόγος που προκλήθηκε αυτό είναι ότι υπάρχει αλλαγή στα, στα των δασών, γιατί πιο πολλά έχουν γίνει κονοφόρα. Αυτό είναι λάθος που πρέπει να πάρουμε πρώτα προχωρήσουμε στο μέλλον. Θα πρέπει η ευρωπαϊκή πολιτική να κάνει σωστή χρήση της κλιματικής αλλαγής. Τι γνωρίζουμε για τα δάση λοιπόν. Ε, τα, η βιοπικιλότητα είναι καλύτερη για το κλίμα γιατί μπορεί να δεσμεύσει μεγάλες ποσότητες ε, ε άνθρακα για εκατοντάδες ετών. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι κατανοητό επίσης. Εξαιτίας της, ε, του πλούτου σε ήδη, η γενετική ποικιλομορφία Θα κάνει πιο ανθεκτικά σε περιβαλλοντικές αλλαγές, κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό υπό το φως της κλιματικής αλλαγής. Τα άσχημα ναι, είναι τη βιοπικιλότητα και τα βιοπικιλά δάση δεν τα πάνε καλά. Έχουμε 2 με 3% μονάχα τις 100 δασών που δεν έχουν ε, ε, πληγή. Η συμβατική λοτόμηση συμβάλλει στην ε, απώλεια βιοπικιλότητας. Έχουμε χάσει ήδη πάνω από 500 ήδη από τα δάση μας και αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί. Σε αυτή τη φωτογραφία βλέπουμε έναν τόπο Natura 2000. Όπως βλέπετε έχει αποψηλωθεί πλήρως. Έτσι προστατεύουμε λοιπόν τα δάση. Και τι συμβαίνει το κλιματικό αντίκτυπο των δασών η καταβόθρα έχει αρχίσει να μειώνεται. Μεταξύ 2009 και 2015 είδαμε μία μείωση της τάξης του 10%. Εκτιμάται ότι στο μέλλον, το 2030, τα επίπεδα συγκομιδής θα αυξηθούν και αυτό θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση ε, στις καταβόφερες θα συνεχιστεί αυτή η τάση και όπως βλέπετε παρόλο που θα υπάρχει λιγότερη αποψήλωση και περισσότερη αναδάσωση, παρόλα αυτά στα συγκεκριμένα δάση οι καταβόθρες τα ε, του Αφρικού θα μειωθούν. Αυτό εξαρτάται και από τις πολιτικές που εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Σε αυτή τη φωτογραφία βλέπετε τι συμβαίνει μετά τη συγκομιδή. Είναι μικρή εικόνα, αλλά το μήνυμα είναι ότι μετά από την ε, συγκομιδή το μισό του άνθρακα χάνεται από το δάσος και χρειάζεται πάρα πολλά χρόνια για να επανακτηθεί αυτή η ποσότητα. Φυσικά έχει και σημασία που χρησιμοποιούμε το ξύλο. Δεν το χρησιμοποιούμε για μακροπρόθεσμα προϊόντα, μόνο το 1 πέμπτο του ξύλου χρησιμοποιείται για προϊόντα ε, που έχουν διάρκεια. Το πιο πολύ το χρησιμοποιούμε για χαρτί, πούλπα και για καύση. Θέλω να δώσω έμφαση στο εξή ότι το κάψιμο των δασών δεν είναι ουδέτερο άνθρακα. Και σίγουρα αυτά τα δέντρα θα είχαν μεγαλύτερη αξία αν τα χρησιμοποιούμε για την ε, δέσμευση άνθρακα στα δάση, αλλά εδώ έχουμε εικόνες από τη Φιλανδία, από τη Γαλλία και από τη Σλοβακία, Σλοβενία, όπου βλέπουμε ότι τα, το ξύλο καίγεται για την παραγωγή ενέργειας. Το 2020 αναμένεται ότι η συνολική συγκομιδή του 2000 30 ε, θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας και θα ε, εκπαιμφθεί στη συνέχεια στην ατμόσφαιρα. Να δούμε τι σημαίνει στην Φιλανδία. Έχουμε μια ενεργική στρατηγική που βασίζεται στο ξύλο ως πηγή ενέργειας και αυτό αναμένεται να μειώσει την καταβόθρα του άνθρακα στα δάση. Η θλιβερή αλήθεια είναι ότι αυτό ε, συμβάλλει στη μεταφορά εκπομπών από τον ένα τομέα στον άλλο. Γιατί παρόλο που θα υπάρξει μείωση εκπομπών, αυτή η μείωση στη ξεμενή του Λουσιεφ θα δείξει ότι δεν θα υπάρχει καθαρή μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030. Άρα θα μπορέσουμε να ε, αμβλύνουμε τις αρνητικές επιπτώσεις και βλέπουμε λοιπόν δεν μπορεί να κάνει κακή εφαρμογή πολιτικής. Η ευρωπαϊκή πολιτική δεν μας ε, φέρνει πιο κοντά στο Παρίσι γιατί για να πετύχουμε τους στόχους χρειαζόμαστε ταχύτατη ε, μείωση των εκπομπών και αρνητικές εκπομπές. Χρειαζόμαστε λοιπόν δάση. Λοιπόν, τι μπορείτε να κάνετε εδώ πέρα. Μπορείτε να να εξασφαλίσετε ότι υπάρξει δράση, να δώσετε οικονομικά κίνητρα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μπορείτε να θέσετε στόχους για το μέλλον και για τις καταβόθρες και να ενισχύσετε την ενεργειακή πολιτική. Επίσης και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και να εφαρμόσουμε επίσης τους νόμους της φύσης. Να πάμε και κάτι θετικό, κλείνοντας, επειδή έχουμε ασφαλή και αποτελεσματικά εργαλεία εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε να υποστηρίξουμε δημιουργία κατά βόθρων, να έχουμε δάση με υψηλή σε άνθρακα, να σταματήσουμε την αποψήλωση. Μπορούμε να έχουμε ε, φυσικές μεθόδους διαχείρισης που έχουν ήδη δοκιμαστεί και να υποστηρίξουμε τη βιοποικιλότητα, να έχουμε χαμηλά επίπεδα συγκομιδής και να ε, εστιάσουμε πιο πολύ σε προϊόντα μεγάλης διάρκειας ε, παράγοντα από ξύλο. Αυτή θα πρέπει να είναι η πολιτική μας. Το τελικό μου slide είναι ότι δεν έχουμε χρόνο, ότι πρέπει να δράσουμε τώρα. Η ατμόσφαιρα νοιάζεται μόνο για τις καθαρές εκπομπές. Ανεξαρτήτου της πηγής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στην κυρία Γιάννη. Thank you very much. Can you hear me? Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε, λέει κυρία Μπακ να σας παρουσιάσω την έκθεση την οποία θα βρείτε εδώ στην αίθουσα αν θέλετε να την πάρετε μαζί σας. Τη συνέταξη του ΕΕΣΑΚ το Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Χάραξη Πολιτικής και στην έκθεση στη σύνταξή της συμμετείχαν 19 εμπειρογνώμονες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες δηλαδή αποτελεί μια επιστημονική προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος της βιωσιμότητας και της πολιτικότητας των ευρωπαϊκών δασών, το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως. Καταρχάς θα σας παρουσιάσω εδώ κάποιες διαφάνειες. η πρώτη με τα κύρια μήνυματά μου και μετά θα πάω σε λεπτομέρειες για να τα διευκρινίσω. Καταρχάς, αναφερόμαστε στο ότι οι χώρες μέλη δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις ε, παγκόσμιες προκλήσεις υποχώρηση βιοποικιλότητας και κλιματική αλλαγή. Οπότε χρειάζεται καθοδήγηση από την Ένωση, κινήτρα και διαφανείς σαφείς πολιτικές ώστε να βοηθήσουμε τις χώρες μέλη στις πολιτικές τους. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι η νομοθεσία για την χρήση υγιής θα πρέπει να είναι σαφής και να μην επιτρέπει μεταφορά ρήπων από άλλους τομείς στην δασοκομεία, ώστε να αποφύγουμε την αύξηση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, το οποίο φαίνεται ότι θα συμβεί αν δεν αλλάξουμε τις πολιτικές που υπάρχουν. Και τέλος, ο πιο αποτελεσματικό τρόπος αποφυγής κινδύνων, όπως το δάσος που ακούσαμε προηγουμένως και για να προωθήσουμε ακριβώς την ανθεκτικότητα και να πετύχουμε τους στόχους βιωσιμότητας είναι το να προωθήσουμε τα ετερογενή δάση τα οποία είναι ανθεκτικά στις διάφορες πιέσεις. Βεβαίως έχουμε και τις φυσικές πιέσεις οι οποίες συμβαίνουν συνεχώς όμως έχουμε εργαλεία για να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Στην έκθεση μας λοιπόν καταγράφουμε κάποιους ε, παράγοντες που αφορούν τα δάση της Ένωσης. Αναγνωρίζουμε δηλαδή ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία στα δάση στην Ευρώπη. Υπάρχουν οικολογικοί παράγοντες, ε, κλιματολογικοί παράγοντες, ε, παράγοντες ανάπτυξης. Έχουμε το θέμα της συγκομιδής. Έχουμε το θέμα της βιώσιμης διαχείρισης των δασών και τους στόχους και το θέμα της βιοποικιλότητας το οποίο δέχεται πιέσεις σε όλες τις χώρες. Επίσης τονίζουμε βεβαίως ότι η δασοκομεία είναι πολύ σημαντικό κλάδος πολλών οικονομιών όπως ήδη ακούσαμε. Και χάρη σε αυτή την αρχή της επικορικότητας οι χώρες μέλη έχουν χαράξει εθνικές δασικές ε, πολιτικές βάσει εθνικών παραδόσεων και όχι έχοντα κατά νου τόσο τι παγκόσμιες προκλήσεις που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η δασοκομεία. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αναπτύξει τρόπους σύζευξη αυτών των εθνικών διαφορών επιτρέποντα ταυτόχρονα στι χώρε να βελτιώσουν την δασική του διαχείριση και να ακολουθήσουν βέβαια και να τηρήσουν τι διαφορετικέ υποχρεώσει του. Όπω λέγαμε προηγουμένω, ότι συμβάλλουν και τα δάση ε, στην κλιματική αλλαγή λόγω αποθήκευση διοξιδίου άνθρακα και ε, τη καταβόθρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε κατά νου για τα δάση μα. Και τέλο, πρέπει να πούμε ότι επανέρχεται ο άνθρακας στην ατμόσφαιρα σε λιγότερο από 10 χρόνια αυτό που συλλέγεται από τα δάση μα. Οπότε εμείς θα πρέπει να θα πρέπει αντί να καίμε τα προϊόντα από τα δάση ή να τα μετατρέπουμε σε χαρτοπολτό, θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά. Και αυτό ακριβώς θα πρέπει να το δούμε σε, ε, στην προοπτική της στρατηγικής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την ε, συγκομιδή η βιοενέργεια είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον και υπάρχει κίνδυνος επιτάχυνσης της κλιματικής αλλαγής εδώ. Η βιοπικιλότητα επίσης βρίσκεται σε υποχώρηση και η σωστή δασική διαχείριση είναι απαραίτητη ακριβώς για να διατηρηθούν οι αξίες της βιοπικιλότητας σε όλο το σχεδιασμό για την ε, διατήρηση αυτών των στόχων της βιοποικιλότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα μπορούσαμε τώρα να λάβουμε υπόψη μας τα δάση όσον αφορά τις πολιτικές αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής στην Ένωση. Υπάρχει ισχυρή όθηση για χρήση βιοενέργειας και προϊόντων της. Αλλά αυτό δεν διασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ της παραγωγής ενέργειας και την ε, διατήρηση του άνθρακα και της πολιτικότητας των δασών. Υπάρχουν βεβαίως διάφορα επίπεδα πίεσης, τα οποία αν παραμένουν στα επίπεδα που είναι, τότε έχουν κίνητρα μεταφοράς ε, ε, ρήπων οι χώρες μέλη, στην δασοκομεία χωρίς ακριβώς δηλαδή να υπάρξει κατάλληλη αντιμετώπιση και στις χειρότερες περιπτώσεις οι χώρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημόσια κονδύλια για να μεταφέρουν ακριβώς ε, ρήπους σε τομείς όπως η χρήση γης, χωρίς πραγματική αύξηση των ρήπων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια πλήρη ισορροπία μεταξύ ε, αποθήκευσης και χρήσης ε, του άνθρακα. Ε, έχουμε δώσει στην εκθεσή μας κάποιες ενδείξεις σε σχέση με την αποθήκευση και του, τα βέλτιστα εργαλεία διαχείρισης, επειδή η διαχείριση δεν είναι ποτέ ουδέτερη όσον αφορά την κλιματική σκοπιά του άνθρακα. Τα καλά νέα είναι ότι η παραγωγή και η διαχείριση των δασών τείνουν να αυξήνουν μακροπρόθεσμα αντί να μειώνουν την ε, παροχή ξυλίας και βοηθούν στη διατήρηση των ε, αξιών της βιοποικιλότητας το οποίο είναι ε, χρήσιμο διπλά. Ας πούμε σε διάφορες χώρες όπου έχουμε κάνει ανάλυση κάποιων δεδομένων, μας δείχνουν οι μελέτες ότι η αποδίκευση του άνθρακα στα υπάρχοντα δάση αποτελεί το φτηνότερο τρόπο, ένα από τους φτηνότερους τρόπους μείωσης των καθαρών ε, ρήπων άνθρακα. Αν έχουμε λοιπόν τη μέσα άνθρακα 10-15 ευρώ το τόνο, ε, αυτή η αποθήκευση θα είναι, πιο, θα, θα είναι βέλτιστη στα δάση παρά αλλού. Τι γίνεται τώρα με τους ιδιοκτήτες δασών και την αποθήκευση. Οικονομικά είναι ένα θετικό στοιχείο και αντίστροφα. Αυτό θα πρέπει να ελέγχεται όμως από παρεμβάσεις στην αγορά, οπότε η, επίδοση, η επιδότηση συγγνώμη, των, της αποθήκευσης άνθρακα αποτελεί το σωστό οικονομικό κίνητρο και θα πρέπει να ακολουθούμε την αρχή ο πληρώνει, το οποίο ήδη εφαρμόζεται και ισχύει στην Νέα και στον Καναδά. Δεν το βλέπουμε όμως να ισχύει αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. η οικονομικά ορθή διαχείριση και η βελτίωση της πολυκληρικότητας. Δεν βασιζόμαστε στη μέγιστη απόδοση, γι' αυτό, αλλά λαμβάνουμε υπόψη μας την πολυλειτουργικότητα και τους ε, κινδύνους κλιματικής αλλαγής. Προτείνουμε λοιπόν στην έκθεσή μας ε, το μείγμα ετερογενών ειδών, ώστε να έχουμε ε, υψηλές υπηρεσίες οικοσυστήματος, ώστε να αντιμετωπίσουμε και τους μελλοντικούς κινδύνους. Σα ευχαριστώ. Μας έμειναν και λίγα λεπτά για συζήτηση. Παρακαλώ ποιοι θέλουν το λόγο. Μπούντα Αγνιού. Κάτεμπαχ. Γιάρ. Close the list and uh, first on my list is Mr. Buddha Florishers. For one minute, please, because we are quite short. Παρακαλώ ένα λεπτό, γιατί μας έμεινε πολύ λίγος χρόνος. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή ε, τις ε, παρουσιάσεις των εμπειρογνωμόνων, αλλά υπάρχουν κάποια κενά. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Ήπεθρο, αλλά στα χωριά ο κόσμος χρησιμοποιεί το ξύλο για θέρμανση. Ε, δεν έχει βρει εναλλακτική λύση από την καύση του ξύλου. Θα στερήσουμε δηλαδή από τον κόσμο ε, τη θέρμαση, γιατί στα χωριά δεν υπάρχει μεγάλη πρόσβαση σε πετρέλαιο. Πρώτα αυτή την, αυτή την απάντηση θα πρέπει να δώσει την ερώτηση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλήσαμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε ολική, ηλιακή και ούτω καθεξής. Γνωρίζουμε τα προβλήματα από τη διαχείριση των δασών. Όλοι θα θέλουμε να διατηρηθούν τα δάση να έχουμε βιώσιμη διαχείριση. Αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε και αλλοδαπές ε, εταιρείε στη Ρουμανία που ε, εκμεταλλεύονται τα δάση μας. Αλλά θα πρέπει να βρούμε εναλλακτική για τη χρήση του καυσόξυλου, για τη θέρμαση. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε στον κόσμο να ζεσταίνεται. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άγνιο, ευχαριστώ. Άκουσα και εγώ τις ομιλίες ε, και αποκόμισα την εντύπωση ότι αν αφήσουμε τα δέντρα στην ησυχία τους θα δεσμεύουν άνθρακα στον αιώνα τον άπαντα. Όταν πεθαίνουν όμως κλείουν και πάλι το, το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ή θα υλοτομούνται και πάλι θα απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και για χαρτοπορτό πάλι σε τελική ανάλυση θα καίγονται και θα απελευθερώνουν πάλι το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ή θα τα χρησιμοποιήσουμε το ξύλο για να κατασκευάζουμε έπιπλα, αλλά και τα έπιπλα μπορούν να καταστραφούν από μικροοργανισμούς, από σαράκια και πάλι καταστρέφονται και πάλι έχουμε απελευθέρωση του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Για να μιλήσουμε για τα εργοστάσια που καίνε, ε, χρησιμοποιούν αυτά τα ξύλα πόσο μπορούν να, παράγουν διοξίδιο του άνθρακα. Και μην ξεχνάτε τον κύκλο όμω. Όσο περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα έχουμε στην ατμόσφαιρα, τόσο πιο γρήγορα θα αναπτύσσονται και τα δέντρα. Σα ευχαριστώ κύριε Κάντεμπαχ. Από τον αδελφό Ένιο απέκλεισε τη δυνατότητα να φτιαχτούν διαμάντια από αυτά τα δέντρα σε γενικέ γραμμέ να σα ευχαριστήσω για την παρουσίαση, τι παρουσίασει που έχουμε εδώ πέρα σήμερα και δείχνει για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει να είμαστε ε, πρόθυμοι να συζητήσουμε διαφορετικά αυτό το θέμα. Γιατί δεν σημαίνει ότι αν έχουμε κάποια δέντρα, αυτά μπορούν να αποτελέσουν ένα καλό δάσος γιατί είναι προπόθεση το δάσο να συμβάλλει στη βιοποικιλότητα και στην προστασία του περιβάλλοντο. και και θα πρέπει επίση να συζητήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε με το προϊόν. Θεωρώ ότι η συνολική συζήτηση για τη βιομάζα είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το για ποια γενιά βιομάζας κάνουμε λόγο. Στην τρίτη παρουσίαση επικράτησε το ερώτημα της κλιματικής αλλαγής. Και φυσικά το ζήτημα αν καίγεται ένα δάσος στο οποίο γίνεται σωστή διαχείριση το ίδιο με ένα το οποίο έχει βασιστεί σε μονοκαλλιέργεια. Και μια πλέον ερώτηση. Σε κάποια σημεία της Ευρώπης ότι χάνονται εκτάσεις ειδικές από την αναδάσωση Δηλαδή επεκτείνονται τα δάση και μειώνονται οι αγροτικές εκτάσεις. Ευχαριστώ. Κύριο Κύριος Γιάρα, ευχαριστώ. Τρεις μικρές παρατηρήσεις όσον αφορά την ε, δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα, δημιουργεί θέσεις για νέα ανάπτυξη ε, την εξολόγηση του, της χρήσης του ξύλου γιατί σίγουρα μπορεί να γίνει σωστή χρήση από, του ξύλου που παράγεται από τους ε, ιδιώτες ιδιώτες ε, δασών. Θα πρέπει να δούμε και τις εναλλακτικέ. Εγώ προτιμάω να και ξύλο παρά με πετρέλαιο. Γι' αυτό θέλω να υπάρξει μια σωστή ταξινόμηση. Υπάρχει είναι σίγουρα καλύτερα να το ανακυκλώσουμε από το να το αφήσουμε και να έχουμε συνέχεια εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. And now... Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα ξαναδώσω το λόγο στις καλεσμένες ε, από τον τρίτο γύρο. Παρακαλώ. Δύο-τρία λεπτά κάθε μία. Ε, καταρχήν ε, να επισημάνω ότι όταν σκεφτόμαστε για την κλιματική δράση για τα δάση και σίγουρα η βιοπικιλότητα είναι υπέρ της κλιματικής λειτουργίας των δασών και αυτό φαίνεται και από τη βιβλιογραφία. Όσο περισσότερη βιοπικιλότητα έχουμε, τόσο πιο ανθεκτικά είναι τα δάση. Είναι αλληλένδετες αυτές οι έννοιες, οπότε μπορούμε να έχουμε μια αμοιβαίως υποφελή κατάσταση. Τώρα, ως προς την ερώτηση τι άλλες εναλλακτικές έχουμε για θέρμανση στα χωριά στην Ήπεθρο. Έχουμε φυσικά εναλλακτικέ ε, λύσεις. Ε, η δυσκολία έγκυται στη διανομή τους. Έχουμε ε, γεωθερμική ενέργεια, έχουμε αντλίες θερμότητας, έχουμε ηλιακή ενέργεια, ολική, αλλά θέλουμε ένα ενεργειακό σύστημα που δεν θα εκπέμπει περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αλλά θα παραμένει το, ο άνθρακας δεσμευμένος σε, σε προϊόντα και στα δάση. Σε ό,τι αφορά το σχόλιο ότι όταν τα δέντρα πεθαίνουν εκπέμπουν άνθρακα, ε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μία χρονική κλίμακα. Το έδειξε και στην τελευταία μου διαφάνεια. 10 με 20 χρόνια μας έχουν μείνει για ουσιαστική, πραγματική πολιτική για, το μετριασμό των των κλιματικών αλλαγών και δυστυχώς στερούμε στην πολιτική μας. Οπότε, αν έχουμε αυτό το χρονικό ορίζοντα 10 με 20 χρόνια, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ξύλο με τέτοιο τρόπο, ώστε σε αυτή την περίοδο να μην δημιουργήσουμε μια πραγματική καταστροφή που θα μας κάνει να, γυρίσουμε, να φτάσουμε σε μια κατάσταση χωρίς επιστροφή, χωρίς δυνατότητα ανάκτησης δηλαδή του κλίματος. Σας ευχαριστώ κυρία Μπέκερ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την σας την Χάνα. Σίγουρα υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις για τη θέρμανση στην Ήπεθρο. δεν είναι μόνο το ξύλο η ενεργειακή και αν συγκρίνουμε τα οικονομικά αποτελέσματα τέτοιων εναλλακτικών λύσεων, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ένα χρονικό ορίζοντα 20 ετίας, 30 ετίας. Θα έχουμε όλο και πιο φθηνούς τρόπους για την παραγωγή θερμότητας και ενέργειας, χάρη σε αυτές τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ηλιακή και άλλες. Θα πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι λοιπόν και να μην ε, επικεντρωθούμε μόνο στον άνθρακα ή στο πετρέλαιο σε εναλλακτική για το ξύλο. Σίγουρα τα δέντρα κάποια στιγμή πεθαίνουν. Αυτό είναι ένα αναφυσβήτητο. Και σίγουρα ε, έχουμε μεγαλύτερη αύξηση ε, του διοξιδίου του άνθρακα σε τέτοια περίπτωση, αλλά αν λάβετε υπόψη στο πλαίσιο των 10-20 χρόνων, όλα τα μόρια άνθρακα που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα θερμαίνουν αυτόματα τον αέρα όπου και αν βρίσκονται στην ατμόσφαιρα. Οπότε αυτό είναι ο κλιματικό αντίκτυπο των εκπομπών. Αν αυτό τον άνθρακα, αυτά τα μόρια τα δεσμεύσουν τα δέντρα, ε, σίγουρα το κάνουν πολύ περισσότερο, για πολύ περισσότερα χρόνια από ότι όταν πεθαίνουν ή όταν κόβονται ή καίγονται. Επίσης, ε, για την βιοενέργεια και τις, τις αμεψισπορές σε γειτονικές των περιοχές που έχουν, έχουν δοκιμαστεί σε πολλές περιπτώσεις ή έχουμε βιοκαύσιμα και ε, βιολογικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις που έχουν ε, ε, ε, που χρειάζονται περισσότερο νερό, περισσότερα θρεπτικά, θρεπτικές ε, ουσίες και τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα είναι πολύ χειρότερα. Οπότε τέτοιου είδους ε, μεθόδους θα πρέπει να τις αναλύσουμε πριν καταλήξουμε στα πραγματικά τους περιβαλλοντικά ωφέλη, αν υπάρχουν. Αυτά και θα ήθελα να κατακλείδη να πω ότι θέλουμε ε, φιλόδοξες εθνικές συνεισφορές ε, και υποσχέσεις ε, προκειμένου να υλοποιήσουμε εμπρόθεσμα τους στόχους των Παρισίων. Και σας παραπέμπω στην έκθεσή μας. Σας ευχαριστώ. Δυστυχώς ο χρόνος μας εξαντλήθηκε, οπότε δεν προλαβαίνω παρά να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εμπειρογνώμονές μας για την ευκαιρία που μας έδωσε να συζητήσουμε αυτό το ε, και πολυστείτε το θέμα της ε, νοσοκομεία και των ε, υπηρεσιών ε, των δασών, υπηρεσιών οικοσυστήματος και υπηρεσιών πρώτη ύλη. Είναι δύσκολη αυτή η ισορροπία και ευελπιστώ ότι θα βρούμε τελικά αυτή την ισορροπία κάποια στιγμή. Ο πρόεδρος Σικέρσκι, να σας υπενθυμίσω ότι η διακομματική ομάδα για τα δάση θα λάβει χώρα ε, στη, στην αίθουσα 5G1 με θέμα αυτή την ε, δασική πολιτική. Και μην ξεχνάτε την ε, χριστουγεννιάτικη μας δεξίωση στο άλλο κτίριο. Αυτά και σας εύχομαι καλό βράδυ.